Bonjour. Καλημέρα. Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Συνάδελφοι, έχω δυστυχώς άσκημα νέα. Μέχρι τις 4 θα προεδρεύω εγώ. Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Διότι η κυρία Κώστα αρρώστησε και δεν μπορεί να έρθει στις Βρυξέλλες σήμερα. <clears throat> Αυτή είναι η κακή είδηση. Ελπίζω να είναι καλύτερα αύριο. Αυτά. Επομένως, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά. Πρακτικά όχι. Ναι. Oui, oui. Vă rog, aveți cuvântul, doamna Ferheane. Ja, ich würde gerne eine Anmerkung zum Protokoll vom letzten Mal machen und bitte darum, diese Anmerkung auch in das jetzige Protokoll. Ένα σχόλιο για τα πρακτικά και θα ήθελα ή δυνατόν να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίας παρατήρησή μου. Γραπτός μάλιστα σας έχω στείλει την παρατήρησή μου, το έχω ήδη υποβάλει στην γραμματεία ως σχόλιο. Όσον αφορά το βραβείο Λούξ, μας μίλησε γι' αυτό η Doris Πακ και νομίζω ότι θα πρέπει και η δική της η παρέμβαση να συμπεριληφθεί στα πρακτικά είχε αναφέρθει σε μια πολύ σημαντική καινοτόμα πρωτοβουλία που από το 2007 έχει κερδίσει ιδιαίτερο κύρος και έγκλη και μπορεί πραγματικά να συμβάλλει πολύ στην πολιτισμική διπλωματία, η κοινοβουλευτική διπλωματία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούν να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι ευρωβουλευτέ στην απονομή του βραβείου Λουξ 2014. Θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα πρέπει στη συνέχεια το βραβείο Λουξ να ενταχθεί περισσότερο στην σφαίρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο βραβείο αυτό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να συμβάλλει βέβαια σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm. Είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και είχαμε πει επίσης ότι θα πρέπει και οι πολίτες να συμβάλλουν περισσότερο, το ευρύτερο κοινό και να δούμε αν υπάρχουν και δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο πρότεινε η κυρία Ντόρι Σπακ, κάτι το οποίο προέκυψε και από τη συζήτηση που ακολούθησε μετά την παρέμβασή τη και θα ήθελε δυνατόν να συμπεριληφθούν, να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα σημεία στα πρακτικά τη προηγούμενη συνεδρίαση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης της 4ης Νοεμβρίου. Δεν υπάρχουν ανακοινώσει του Προέδρου. Έχουμε δερμηνία στα αγγλικά, γαλλικά, δανέζικα, εστονικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και ελληνικά. Κύριε Μπλάχαϊμα, πρότεινε να μας μιλήσει για το Internet Governance Forum, Φόρουμ Διακυβέρνησης του Ίντερνετ. Σας, ευχαριστώ συνάδελφοι. Συμμετείχα στην προηγούμενη συνεδρίαση του φόρουμ όσον αφορά τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και θα ήθελα απλώς να κάνω ένα σύντομο απολογισμό της συζήτησης αυτής που διεξήχθη. Έχουμε ηλεκτρονικά επίσης και κάποιες παρατηρήσεις της Επιτροπής ΙΤΡΕ. Ε, Θα ήθελα να αφαιρθώ απλώς σε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ε, σχέση με τη δική μας την Επιτροπή. Το Internet Governance Forum, το Φόρουμ Διακυβέρνησης του Διαδικτύου, ήδη φύσταται εδώ και 9 χρόνια. Ξεκίνησε στην ε, Τίνιδα, στα πλαίσια του Φόρουμ Συμμετοχής Κυβερνήσεων Εταιριών πολιτών, όπου είπαμε λοιπόν στην Τίνιδα ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πολυμερές φόρουμ όπου να συμμετέχουν διάφοροι εμπλεκόμενοι, ενδιαφερόμενοι. Ένα στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς όλος ιδιαίτερος είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε net neutrality, η ουδετερότητα δηλαδή στα πλαίσια του διαδικτύου. Νομίζω το ζήτημα είναι πολύ ενδιαφέρον και από ευρωπαϊκής και από παγκόσμιας πλευράς και το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδίω για τι αναδυόμενε χώρε, γιατί ορισμένε εταιρείε, ορισμένε επιχειρήσει παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μόνο όμω για συγκεκριμένο περιεχόμενο, για παράδειγμα για συγκεκριμένε ιστοσελίδε ή για το Facebook. Και συνειδητοποιείται ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη συζήτηση που διεξάγεται και στι χώρε αυτέ, αλλά και τη συζήτηση που πρέπει εμεί να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο, να καταφέρουμε να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που έχουμε ήδη εντοπίσει εμείς εδώ στην Ευρώπη, να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ενσωματώσουμε πολυμερείς μηχανισμούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο θίξαμε ήταν η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε εξαιτία τη δική μα θεωρώ συμβολή ε, στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη είναι η προστασία των παιδιών online. Ξέρετε το ζήτημα αυτό μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Έχουμε κάνει πολύ έντονες συζητήσεις για το ζήτημα αυτό. Η όλη συζήτηση που κάναμε στα πλαίσια της, ε, του Φόρουμ για την Κυβέρνηση του Διαδικτύου κατέληξε συμπέρασμα ότι θα πρέπει όλο και περισσότερο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμβάλλουν περισσότερο στο να δημιουργήσουμε ένα διαδίκτυο το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές ιδίω για τους ανήλικους, ιδίω για τα παιδιά. Πιστεύω λοιπόν ότι από κοινού εμείς ως Ευρωπαίοι με τους άλλους εταίρους μας εκτός Ευρώπης θα μπορούσαμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Συστήσαμε επίσης το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με την Τουρκία, Δυστυχώς στην χώρα αυτή και ιδίω στην Κωνσταντινούπολη φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να διοργανωθεί το φόρουμ αυτό. Γίνανε μάλιστα διάφορες προσπάθειες προκειμένου να μποϊκοτάρουν το φόρουμ αυτό. Θελήσανε να προωθήσουν ένα διαφορετικό φόρουμ και αυτό πιστεύω είναι πραγματικά κρίμα γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την Τουρκία και τα οποία θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί στα πλαίσια ενό τέτοιου φόρουμ όπω η ελευθερία έκφραση και το καθεξή. Ελπίζω ότι στο επόμενο φόρουμ που θα γίνει στην Βραζιλία θα είμαστε θέση να αναφερθούμε περισσότερο στα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα δηλαδή του διαδικτυακού πλουραλισμού, να ενταχθούν στα πλαίσια αυτού του φόρουμ και όχι στα πλαίσια κάποιου άλλου ανταγωνιστικού φόρουμ. Τώρα, το 2015 είναι ουσιαστικά το τελευταίο έτος διοργάνωσης του φόρουμ αυτού. Τα Ηνωμένα Έθνη θα αποφασίσουν αν η εντολή του φόρουμ αυτού θα ενισχυθεί, αν θα παραταθεί και θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλες συνεδράσεις μετά το 2015. Πρέπει να βρεθούν βέβαια κάποιες συγκεκριμένε τεχνικές λύσεις όπως η χρηματοδότηση της γραμματείας του φόρουμ αυτού. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα δοθεί, πιστεύω, μεγαλύτερη προβολή στο φόρουμ αυτό, αλλά προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να προσληφθεί και περισσότερο προσωπικό, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή το φόρουμ αυτό βασίζεται μόνο στην γραμματεία που έχει στα πλαίσια των Εθνών, η οποία απασχολεί ελάχιστου εργαζομένου. Συστήσαμε επίσης το ζήτημα του ICANN καθώς επίσης και το ζήτημα της ε, λογοδοσίας του ICAN, και αν θα μπορούσε να ενταχθεί στη διαδικασία Ριάδνη. Θελήσαμε να δούμε αν ε, μπορούμε να διεθνοποιήσουμε κάπως το ζήτημα της ευθύνη, της λογοδοσίας και της διακυβέρνησης του διαδικτύου, χωρίς οι σημαντικές αυτές αποφάσεις να λαμβάνονται αναγκαστικά από κάποιους ορισμένους μονοπαράγοντες μεμονωμένα. Τώρα όσον αφορά τα έγγραφα τα οποία θα λάβετε θα δείτε τις διμερείς επαφές τις οποίες είχαμε. Είχαμε κάποιες έντονες συζητήσεις με νέους στα πλαίσια του Φόρουμ Νεολαίας, του Youth Forum. Συζήτησαμε για τις ανάγκες των νέων και για τη δική του την άποψη όσον αφορά τα ευαίσθητα ζητήματα στα πλαίσια της διακυβέρνησης του διαδικτύου. Σας καλώ να διαβάσετε τα έγγραφα αυτά και τα πρακτικά που είχαμε από τη συνεδρίαση και από τις άλλες επαφές που είχαμε στα πλαίσια του φόρουμ. Αποφασίσαμε να συμμετάσχουν δύο εκπρόσωποι από την Επιτροπή Πολιτισμού στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει του χρόνου και κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε πίσω περισσότερες πληροφορίες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είμαστε θέσει να συνημερώσουμε πολύ καλύτερα κατά αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω πάντως ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης αλλά και άλλα ευρωπαϊκά φόρουμ θα πρέπει να συμβάλλουν στο να προβληθεί πολύ περισσότερο το φόρουμ αυτό για την βέλτιστη διαχείριση του διαδικτύου. Θέλω να ελπίζω ότι του χρόνου θα έχουμε και εκπροσώπους από την Μεγάλη Βρετανία. Ελπίζω ότι θα έχουμε και Βρετανούς ευρωβουλευτές, αλλά θα πρέπει να έχουμε και εκπροσώπηση από άλλες χώρες, καθότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω της πολυμερούς αυτής προσέγγισης να προωθήσουμε περισσότερο τις βασικές αυτές αρχές διαχείρισης του διαδικτύου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 έκανε η συνάδελφο. Εάν όχι, θα περάσω το επόμενο θέμα, απαλλαγή 2013, Γενικός προπολογισμό Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Νοέμβριο η, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μια έκθεση όσον αφορά τον προϋπολογισμό του προηγουμένου έτους και πρέπει να εγκρίνει την όλη διαχείριση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα τα θεσμικά όργανα. Στις 5 Νοεμβρίου το ελεγκτικό συνέδριο παρουσίασε την εκθεσή της για το 2013, την οικονομική εκθεσή της. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών μελέτησε την εκθεσή αυτή και κάθε μία από τις ε, επιτροπές πρέπει να γνωμοδοτήσει. Ο δικός μας συνάδελφος της τάξης της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Φερνάντο Μάουρα Μπαρανταριάν. Πρέπει να είναι έτοιμη η γνωμοδότησή μας στις 12 Ιανουαρίου η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 9η Δοκέμβριου. Σας δίνω το λόγο, αγαπητέ συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, σήμερα θα σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας μέρος της Επιτροπής εκ μέρους των προπολογισμών που είναι επί της ουσίας υπεύθυνη. Πρόκειται για θέματα που αφορούν για το 2013 την βασική προτεραιότητα. Η απαλλαγή θα πρέπει να γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συγκεκριμένο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρουσιάζουμε λοιπόν εδώ την πολιτική πτυχή του ελέγχου που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον έλεγχο επί του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόψη αυτή βασίζεται στην θεώρηση πρώτα απ' όλα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του 2013 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Οπτικοαστικών Μεθεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, την ε, ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και η πρόταση, στην πρόταση ψηφίσματος προτείνω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, είναι θετικό αυτό το οποίο λέγεται για προετεραιότητα όσον αφορά τα προγράμματα ανελίσσες και εράσμους Plus. Δεύτερον, με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό εκτέλεσης για τα προγράμματα έως το 2013, 2007-2013, για την νεολαία σε δράση, για τους τομείς, και για τους τομείς πολιτισμού και μέσων ερισμένωσης εκτελέστηκαν σε ποσοστό 100%. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που εγκρίθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια αρνητική κατάσταση το επόμενο έτος. Δεν θα θέλαμε αυτή η κατάσταση να επαναληφθεί στα νέα προγράμματα. Τρίτον, διαπιστώνουμε ότι ο εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης οπτικουστικών θεμάτων και πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΑΘΕ όπως ονομάζεται, εκτέλεσε το 96% των πληρωμών του εντός των συμβατικών χρονικών ορίων. Και θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν άμεσες επιπτώσεις στα δικαιώματα των δικαιούχων και θα ήθελα να ενθαρρύνω τον εκτελεστικό αυτό οργανισμό να βελτιώσει τα συστήματα ελέγχου που διαθέτει. Τέταρτον, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας οργάνωσε πολλές δραστηριότητες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών. Συγχρόνως, είπαμε ότι ήταν επίγουσα ανάγκη η προετοιμασία για τις περικοπές που θα γίνουν στο προπολογισμό του 2014 ναι. για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Σήμερα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, την οποία ήμουν και εγώ εισηγητής, είναι ο μοναδικός και άμεσος σύνδεσμος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών Παρ' όλα αυτά, το επίπεδο χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά χαμηλό και θα πρέπει να εμπλουτιστεί και το περιεχόμενό του με νέες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να πω ότι είμαι αντίθετος προς οποιοδήποτε περαιτέρω περικοπή του προγράμματος η Ευρώπη για τους πολίτες για την χρονική περίοδο 2014-2020. Αυτή είναι η έκθεση που ήθελα να σας παρουσιάσω και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μάουρε. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Δεν είναι κανείς εδώ. Ε, κυρία Μπίργκετ, μήπως θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Μαρτίν Cineva dintre deputați? Μεταξύ των συναδέλφων θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο κάποιος. Θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επεσήμενο ο εισηγητής ότι είναι ο αντίθετος σε οποιαδήποτε ε, περικοπή στα πλαίσια του προγράμματος που προβλέπεται για τους πολίτες τη Ευρώπη 2014 2014-2020. Ήθελα να ξέρω για φέτο, αν μπορεί να μας πει η Επιτροπή εάν υπάρχουν προβλήματα στην ε, καταβολή κονδυλίων για τα προγράμματα στα πλαίσια των δυσκολιών για τον προπολογισμό και στα πλαίσια του διορθωτικού σχεδίου προπολογισμού. Πες μας εσείς πώς εφαρμόζεται εδώ ο προπολογισμό στα πλαίσια του κομματιού αυτού και των προγραμμάτων που αφορούν την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Οργανό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον συντάκτη γνωμοδότησης, τον κύριο Μάουρα Μπαραντιεράν, για το εξαιρετικό σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο μας παρουσίασε είναι ιδιαίτερα ευσύνοπτο το κείμενο αυτό, παρόλα αυτά όμως κατάφερε να τονίσει όλα τα σημαντικά αυτά στοιχεία που έχουν να κάνουν με, τον, με την απαλλαγή όσον αφορά τον προπολογισμό για το οικονομικό έτος 2013. Συμφωνώ ότι η ετήσια αυτή διαδικασία απαλλαγής δεν είναι απλώς μία συνηθισμένη διαδικασία χωρίς ε, ουσία, χωρίς νόημα. Νομίζω ότι αντίθετα δίνει τη δυνατότητα σε εμά, τους ευρωβουλευτές, να μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε πώς εφαρμόζονται εμπράκτος οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το προπολογισμό. Ξέρετε ότι ε, σύμφωνα με τη συνθήκη εμείς μπορούμε να δώσουμε την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δούμε πρώτα ότι οι λογαριασμοί έχουν εφαρμοστεί, έχουν εκτελεστεί σωστά. Αλλά πέρα από το αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγχουμε επίσης και την ίδια την ποιότητα των ε, προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή κάθε φορά να βλέπουμε τα προγράμματα αντιστοιχούν οι στόχου που έχουμε θέσει. Σε μια τόσο δεινή περίοδο από οικονομική πλευρά, πάρα πολλοί πολίτε σε πάρα πολλέ χώρε καλούνται να κάνουν τεράστιε θυσίε προκειμένου οι χώρε του να μπορούν να έχουν ισοσκελισμένου προπολογισμού. Καλούμεθα λοιπόν και εμεί ω Ευρωβουλευτέ να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και να δούμε αν πραγματικά ο κοινοτικό προπολογισμό όντω αντιστοιχεί σε κάποιου συγκεκριμένου στρατηγικού στόχου Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν η χρηματοδότηση αυτή πραγματικά έχει οδηγήσει σε μια ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επί τη ουσία, όπω πολύ σωστά είπε και ο συντάκτη γνωμοδότηση, δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα λογιστικά για το 2013 όσον αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων της αρμοδιότητας της δικής μας της Επιτροπής Διαβίου Μάθηση, Νεολαία Ενδράση και Εκπαίδευση. Θεωρώ ότι οι λογαριασμοί πραγματικά έχουν ε, εκτελεστεί σωστά σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες και δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό ουσιαστικό σφάλμα στους λογαριασμούς αυτούς. Βλέπουμε ότι ορισμένες φορές έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα, κυρίως στα προγράμματα εκείνα, τα περιφερειακά ή στα προγράμματα μεταφορών, η ανάπτυξη πέθρου, όπου έχουμε συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα την περίοδο 2007-2013, το 2013 είδαμε ένα υψηλό επίπεδο υποεκτέλεσης συγκεκριμένων προγραμμάτων. Από την άλλη καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα που είχαν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου όταν μας παρουσίασε την ετήσια έκθεση του 2013, ο προπολογισμό του 2013 χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αιμονή στον τομέα των δαπανών, ενώ θα έπρεπε να μας είχε αποσχολήσει περισσότερο η ποιότητα των προγραμμάτων ή η δυνατότητα εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. Μπορούμε εν γέννη πάντως να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προπολογισμού του 2013. Είδαμε ότι το 2013 στα πλαίσια του προγράμματος διαβίου μάθησης υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση όπου είχαμε τρία εκατομμύρια παιδιά τα οποία θέλει να αποφεληθούν του προγράμματος αυτού, πρόγραμμα το οποίο προβλέπει κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη. Όσον αφορά το πρόγραμμα το οποίο έχουμε στη γραμμή προπολογισμού 399, βλέπουμε ότι εδώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εθνικοί προπολογισμοί που έχουν ως στόχο την αξιοποίηση του της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μειώνονται, παρουσιάζουν πάρα πολύ σημαντική μείωση. Θεωρώ ότι στόχος μας θα πρέπει είναι να αντιστρέψουμε την τάση αυτή και πραγματικά δεν θα πρέπει να απογοητεύσουμε τους νέους οι οποίοι περιμένουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα από την Ευρώπη. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές ανησυχούμε ιδιαίτερα εξαιτία των περικοπών αυτών που έχουμε εντοπίσει όπως σας είπα στον τομέα του πολιτισμού. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσουμε ακόμα περισσότερο στη γνωμοδότηση αυτή ότι ε, στα τέλη του προηγούμενου έτους υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες πληρωμών και τις πιστώσεις πληρωμών, τα διαθέσιμα δηλαδή κονδύλια προκειμένου να εκτελεστούν συγκεκριμένα προγράμματα. Νομίζω ότι η τάση αυτή συνεχίζεται και στο τρέχον, ε, τρέχον με συγχωρητέτος του 2014 και θεωρώ ότι πρέπει να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό γιατί βάλεται η ίδια η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα στα οποία αναφερόμαστε είναι θεμελιώδους σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, προγράμματα όπως το Erasmus Plus και Καταλαβαίνετε ότι αν δεν καταφέρνουμε να αποκριθούμε στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε για τα προγράμματα αυτά, ουσιαστικά έχουμε νέους ή, οικογένει, τις οικογένειές τους οι οποίες δεν καταφέρνουν τελικά να έχουν τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά, προγράμματα τα οποία εντάσσονται στο Erasmus Plus. Θεωρώ ότι και ο συντάκτη γνωμοδότηση, καθώ επίση και οι σκιώδει εισηγητέ από τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε, θα συμφωνήσουν με τι επιπλέον αυτέ παρατηρήσει μου και θα καταφέρουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα συνενετικό συμβαστικό κείμενο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Συμφωνώ με τις, προ... με τις προτάσεις του. Για το 2013 διαπιστώνουμε ότι για όλα τα προγράμματα που αφορούν εμάς, που είναι δική μας δικαιοδοσία, είναι όλα επιτυχή και έχουν εκτελεστεί κατά 100% πράγμα που δεν μπορούμε να το πούμε για όλα τα άλλα προγράμματα της Ένωσης. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι για το 13 και ευχαριστώ εδώ και η Δημιόλγα Τρούπελ για αυτά που είπε το 14 εκ νέου θα διαπιστώσουμε ότι δεν εξισώνονται, δεν ισορροπούνται οι δεσμεύσεις με τις πληρωμές. Αυτό δεν οφείλεται σε εμά, αλλά στο Συμβούλιο που δεν μας χορήγησε τα ποσά που χρειαζόμασταν. έτσι ώστε μεταξύ άλλων οι νέοι που ενδιαφέρουν αυτά τα προγράμματα να μπορούν να έχουν τους πόρους που χρειάζονται για τις διαμονές τους στο εξωτερικό, σε χώρες εκτός από τη δική τους. Εφόσον όμως, αυτό είναι σκάνδαλο γιατί εφόσον έχουν εγκριθεί προγράμματα πρέπει και να πληρώνονται. Ευχαριστώ κύριε Μαρκάνο για αυτά που είπατε και νομίζω ότι πρέπει αυτό να τονιστεί κι άλλο στην έκθεση, ότι ως κοινοβούλιο δεν είμαστε πια διατεθειμένοι να δεχτούμε τέτοια πράγματα, αυτό το παιχνιδάκι του Συμβουλίου που μας το κάνει κάθε χρόνο, ιδιαίτερα για θέματα παιδείας που ενδιαφέρουν τους νέους. Γιατί έτσι χάνεται αξιοπιστία των νέων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνοι δεν ξέρουν αν φταίει το Κοινοβούλιο ή η Κομισιόν ή το Συμβούλιο, λένε η Ευρώπη φταίει. Ενώ εδώ το πρόβλημα είναι του Συμβουλίου, αυτό δύσκολα εξηγείται. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πούμε ρητότερα στην έκθεση. Θα παρακαλούσα δε την Κομισιόν να μας πει για το 14 τι συμβαίνει με τις πληρωμές. Ποιος είναι ο ρυθμός πληρωμών για το έρασμος και άλλα προγράμματα που ενδιαφέρουν τους νέους. Θα ήθελα να επανέλθω στο Έρασμος ΣΥΝ και το προηγούμενο, το παλιό πρόγραμμα Έρασμος. Γιατί το θέμα που τίθεται δεν είναι μόνο τι ποσά εγκρίνει το Συμβούλιο, αλλά πιο συγκεκριμένα πώς μεταφέρονται και εφαρμόζονται όλα αυτά. Μπορεί ένα πανεπιστήμιο να ζητήσει για χι αριθμό φοιτητών πρόγραμμα έρασμος και μετά να διαπιστωθεί ότι είναι λιγότεροι φοιτητές από ό,τι προβλέπονταν και να λάβει λιγότερα ή το αντίθετο. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια ασάφεια στο σχεδιασμό που δείχνει ότι άλλα συζητάμε εδώ και άλλα μπορούν να διαπιστωθούν επί για το θέμα λοιπόν της μεταφοράς, όπως θα πούμε και στο σημείο 6 του νέου έρασμος συν από το 14 και μετά, πρέπει να προσέξουμε τα προγράμματα να μπορούν να εφαρμοστούν. Βέβαια είναι προγράμματα που τα εκτιμούν ιδιαίτερα οι νέοι και όχι μόνο οι νέοι όλο το πρόγραμμα στο σύνολό του το εκτιμούν όλοι. και μη φοιτητέ. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουμε, γιατί με αυτού του είδους τα προγράμματα μπορούμε να πληροφορήσουμε καλύτερα τον κόσμο για αυτό που είναι η Ευρώπη. Δεν είναι μόνο καθαρά οικονομικά προγράμματα, αλλά και επικοινωνιακά και σύνδεσης και σχέσεις με τους πολίτες. Αυτά έλεγε πάντα και η Δωρής Πακ. αυτό που είναι κρίμα και το τονίζω εδώ είναι ότι δεν καταφέραμε τα κράτη-μέλη όλα μαζί στα πλαίσια του προγράμματος για την Ευρώπη των πολιτών να δεν κατάφεραν να, να αποφασίσουν για τον προπολογισμό ενώ πρόκειται για ποσά που δεν είναι τεράστια νομίζω ότι είναι στοιχειώδη μέσα που τα χρειαζόμαστε και που δεν, δεν έχουν τεράστια επίπτωση στον προπολογισμό. Και παρόλα αυτά μειώνονται κατά ένα τέταρτο. Όταν λέμε ότι θέλουμε ο πολίτης να δέχεται πιο εύκολα την πληροφόρηση για την Ευρώπη πρέπει και να το κάνουμε. Χαίρομαι που η συγκητής το τόνισε αυτό. Και δεν ισχύει μόνο για το παρελθόν αλλά και για τα μελλοντικά προγράμματα. Πρέπει να φροντίσουμε όταν υπάρχουν προγράμματα που δεν αποφέρουν κέρδος αλλά που έχουν άλλο είδους όφελος για το κύρος και την αξιοπιστία της Ευρώπης να μην κάνουμε το αντίθετο από αυτό που στοχεύουμε. Ίσως μπορεί να μας πει και η Κομισιόν τα κράτη-μέλη στη συζήτηση στο Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό ίσως να είπανε γιατί να περάσουμε από το ενωσιακό επίπεδο κατευθείαν στα κράτη-μέλη. Ναι, αλλά δεν έχουν κανένα λάβει καμία άμεση δέσμευση τα κράτη-μέλη για προγράμματα για τους νέους και ανταλλαγές κλπ. Αν λοιπόν περικοπεί ο προϋπολογισμός στο ενωσιακό επίπεδο τότε πρέπει να αντισταθμίζεται αυτό εθνικά. Εγώ δέχομαι να γίνει αυτή η αλλαγή αλλά με τον όρο αυτόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος το Νομίζω ότι η γνωμοδότηση ήταν πάρα πολύ καλή και κέρια και επεσήμανε ορισμένα βασικά ζητήματα. Το κυριότερο αυτό είναι αυτό που έδειξε η συνάδελφος Πέτρα, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμές και για προγράμματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε χώρες που υφίστανται μια αδεινή οικονομική κρίση όπως η Ελλάδα και όπου η ανεργία και τα προβλήματα των νέων έχουν ξεπεράσει κάθε όριο τουλάχιστον η αξιοπιστία στις πληρωμές είναι βασικό γεγονός. Λυπούμε όμως αλλά πρέπει να κάνουμε μια γενικότερη παρατήρηση. Ενώ ακούει κανείς ε, από την Κομισιόν και από άλλους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλα λόγια για τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό που είναι και αληθινά ότι αυτά είναι τα θεμέλια της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα με τις περικοπές των προϋπολογισμών, με την απίστευτη γραφειοκρατία αλλά και με τις καθυστερήσεις πληρωμών η εικόνα που δίνουν θα έλεγα τα ανώτερα κλιμάκια της Κομισιόν είναι ότι τον πολιτισμό τον έχουν μόνο για να διαφημίζουν λιγάκι τον εαυτό τους και πολύ λίγο για να του δώσουν πρακτική σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ από την Επιτροπή, κυρία Μπριζίτ Ντοβός. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το σχέδιο ε, γνωμοδότησης ε, του συναδέλφου σας. Θα το λάβουμε υπόψη και θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή πραγματικά προσδίδει μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό των ε, πιστώσεων πληρωμών για τα προγράμματα αυτά. Προσπαθούμε στα μέτρα του δυνατού να αποφύγουμε αρνητικές επιπτώσεις με κυρίως για τους δικαιούχους. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να σας τις αποστείλουμε γραπτός Δεδομένου ότι σήμερα δεν εξετάζεται η απαλλαγή, μπορούμε όμως να σας τις στείλουμε γραπτός. Ο συνάδελφος που ασχολείται με αυτό το θέμα μπορεί να σας πει περισσότερα πράγματα στο σημείο 6 που αφορά περισσότερο το πρόγραμμα Erasmus Plus. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο Φερνάντο Μάουρα, τον συντάξη γνωμοδότησης, να απαντήσει τα σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, αρχίζοντας, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλια που έκαναν σε σχέση με την ε, απαλλαγή. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα να είναι η έκθεσή μου αυτή μια έκθεση που μόνο θα έκανε αξιολόγηση του προγράμματος. Αυτή ήταν η υποχρέωσή μου σήμερα το απόγευμα, αλλά παρόλα αυτά θέλησα να εισαγάγω και κάποια σημαντικά άλλα στοιχεία που με απασχολούν που απασχολούν όλους σε σχέση με το μέλλον. Και παρατηρώ ότι και εσείς συνάδελφοι αναφέρεστε στα ίδια θέματα αυτά που ανέφερα κι εγώ. Κάποιες από τις ε, εκφράσεις και τα σχόλια που άκουσα από τους συναδέλφους, δηλαδή το ότι τα προγράμματα αυτά δεν είναι απλώς προγράμματα τεχνικής φύσεως, τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε από την οικονομική πλευρά. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι ποιοτικά, αν θέλετε, η ψυχή της Ευρώπης, όπως ελέγχθη σήμερα το απόγευμα. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι πρέπει να καταθέσετε όσες τροπολογίες πιστεύετε ότι πρέπει να καταθέσετε και να είστε βέβαιοι ότι στο πλαίσιο του δυνατού θα τις συμπεριλάβω στην τελική μου γνωμοδότησα, δεδομένου ότι πιστεύω ότι εμπλουτίζουν με ουσιαστικό τρόπο την ε, έκθεση που παρουσίασα σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Τώρα θα δώσω στην ε, κυρία Μπόσκος για να συνεχίσει με την Προεδρία. Ελπίζω ότι είναι ξεκούραστη. Ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα μας είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους βραβευθέντες του ευρωπαϊκού βραβείου Καρλομάγνου για την νεολαία 2014, το οποίο εσπίστηκε από το 2008 με στόχο να ενθαρρύνει την δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των νέων για να συμμετέχουν σε προγράμματα ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και απονέμεται σε νέους οι οποίοι ε, προαγάγουν την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και θέλουν να προαγούν και την ε, σύνολο των πολιτών της Ευρώπης που ζουν μαζί. Κάθε χρόνο απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Ίδρυμα ε, με το Ίδρυμα Κάρλο Μάγρου που βρίσκεται στο Άχεν. Πρώτο βραβείο 5.000, δεύτερο 3.000, δεύτερο, τρίτο δεύτερο και οι νικητές καλούνται στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και οι εκπρόσωποι των 28 εθνικών σχεδίων θα κληθούν στο Άχεν σε ένα βραβείο τεσσάρων ημερών. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα τους ε, δώσει το βραβείο και κάποιος εκπρόσωπος από το Ίδρυμα Καρλομάγνου του Άχεν. Σήμερα χαιρετίζουμε στην ε, συνάντησή μας τέσσερις εκπροσώπους την ομάδα που νίκησε, το πρόγραμμα που κέρδισε είναι Our Europe. Αυτό είναι το πρώτο βραβείο. Το δεύτερο πάει στην Iris Pass και στον Kevin Van Dalen από το Young Telephone Coven. Το τρίτο, Employment for You, με εκπροσώπους από την Κύπρο, την ε, Ευανθία Μπογιάζη και τη Χριστίνα και θα δώσω το λόγο σε κάθε ομάδα για 10 λεπτά και μετά θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και πρέπει να πω ότι θα πρέπει από τις ε, 5 και 4 και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά τα θέματα και θα μας κάνει και μια παρέμβαση το Erasmus Plus. Παρακαλώ λοιπόν ο καθένας να σεβαστεί το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αρχίζουμε λοιπόν με τους πρώτους νικητές. Ο Πίτερ ή η Έλενα, ποιος από τους δύο. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το 2011 είχαμε την ιδέα να διασχίσουμε την Ευρώπη, να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για να συναντήσουμε νέους σαν και εμάς. Το 2011 η Ευρώπη είχε πάρα πολλά προβλήματα και μας ενδιαφέραν τα προβλήματα αυτά. Εξοικονομήσαμε λοιπόν χρήματα για δύο ολόκληρα χρόνια γιατί θέλαμε με ή άνευ χρηματοδότηση να μας ενθέσει να κάνουμε το ταξίδι αυτό, το οποίο διήρκησε τελικά μέχρι το Μάιο του 2014. Και έτσι εμείς με τον Πίτερ και την Ελένα πήγαμε σε 24 ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια ενός μεγάλου διπορικού. Συναντήσαμε πάρα πολλούς Ευρωπαίους και μάλιστα μείναμε και στα σπίτια ορισμένων από αυτούς. Βλέπετε εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες από το ταξίδι ενώ όσο ταξιδεύαμε κοινοποιούσαμε στην ιστοσελίδα μας αυτή διάφορα σύντομα άρθρα, βίντεο, ραδιοφωνικά προγράμματα. Βλέπετε μία εκδοχή στα δανέζικα και μία στα αγγλικά. Και ουσιαστικά δημιουργήσαμε αυτές τις μικρές ιστορίες προκειμένου να κοινοποιήσουμε προς τα έξω όλα αυτά τα οποία βλέπαμε επιτόπου στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρήσαμε ότι αν πραγματικά πρέπει εμείς εκ πρώτης όψεως μάλλον από πρώτο χέρι να καταφέρουμε να μάθουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, πώς είναι η κατάσταση των νέων σε διάφορες χώρες, θεωρήσαμε ότι αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όλους τους νέους παντού στην Ευρώπη και μάλιστα 21 σχολεία από τη Δανία μας παρακολουθούσαν μέσω Skype και κάθε εβδομάδα προσπαθούσαμε να έχουμε μία τηλεδιάσκεψη με ένα σχολείο της Δανίας προκειμένου να ενημερώνουμε κάθε φορά μαθητές από τη Δανία για το πού είμαστε, ποιους συναντάμε και ποια είναι τα βασικά μελήματα, οι βασικές ανησυχίες των Ευρωπαίων που συναντούμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε πάνω από 2.000 μαθητές από τη Δανία. Μπορούσαν λοιπόν και αυτοί μέσω του Skype να ενημερωθούν για την κατάσταση των συνομιλικών τους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το σχέδιο αυτό συνεχίστηκε και αφού επιστρέψαμε στη Δανία πριν από 6 μήνες, διότι ε, πάλι εμείς οι δύο έχουμε δώσει 50 διαλέξεις σε διαφορετικά σχολεία, συνολικά σε 8.000 μαθητές από τη Δανία και από άλλες χώρες οι οποίοι φοιτούν στη Δανία. Μοιραστήκαμε λοιπόν μαζί τους διάφορες φωτογραφίες και διάφορα βίντεο από το ταξίδι μας αυτό και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν οι μαθητές πραγματικά να έχουν μια πολύ ζωντανή άποψη, μια πολύ ζωντανή εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα στην Ευρώπη για πάρα πολλούς νέους. Βλέπουμε επίσης ε, μέσω των ε, βίντεο αυτών ε, διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους νέους όπως η άνοδος της ακροδεξιάς, οι ακραίες τάσεις, η ανεργία των νέων κτλ. Μπορέσαμε επίσης να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον πάρα πολλών νέων, να εμπνεύσουμε τους νέους προκειμένου να συνεχίσουν την όλη αυτή συζήτηση και προκειμένου να μιλήσουν όλο περισσότερο για το ζήτημα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Επικεντρωθήκαμε στα πλαίσια του project αυτού, όπως σας είπα, στους νέους της Ευρώπης. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν πάρα πολύ θετικό από την σκοπιά των νέων να καταφέρουμε να τονίσουμε όλες αυτές τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές της κατάστασης των νέων όπως αυτές εμφανίζονται σε διάφορες χώρες. Έχουμε πλέον δημιουργήσει ένα τεράστιο ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό δίκτυο. Είμαστε σε επαφή με 200 τουλάχιστον από τους νέους που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια του διπορικού μας. Και αυτή τη στιγμή καταπιανόμαστε με ένα νέο project, το οποίο θέλουμε να κάνουμε πάλι, και μετά από τρεις ή τέσσερις μήνες πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να έχουμε ετοιμάσει και ένα ντοκιμαντέρ μέσω του οποίου θα εκθέτουμε περισσότερο την κατάσταση των νέων με τη συμμετοχή περισσότερων νέων αυτή τη φορά από περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε αν θέλετε ένα μέσο έκφρασης για πάρα πολλούς νέους στην Ευρώπη και θα μπορούσαν και άλλοι να εμπνευστούν από το δικό μας το παράδειγμα και να αναλάβουν δράση. Αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, Ο βασικό λόγο για τον οποίο προχωρήσαμε στο project αυτό ήταν ότι θέλαμε να καλύψουμε βασικά ποιοι είναι οι συνομιλικοί μα στην Ευρώπη. Είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, οι νέοι που πολύ συχνά του αποκαλούμε η χαμένη γενιά. Θέλαμε λοιπόν να δούμε στην πράξη πώ έχουν τα πράγματα. Ξέρετε ότι πολύ συχνά έχουμε κυρίω εμπειρογνώμονε, πολιτικού, δημοσιογράφου, οι οποίοι παίρνουν το λόγο και οι οποίοι τελικά καταλήγουν συμπεράσματα για το πώ είναι η ζωή των νέων σήμερα. Θεωρήσαμε εμεί ότι θα έπρεπε να δώσουμε, αν θέλετε, φωνή περισσότερο, να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ, ένα βήμα για να καταφέρουν να εκφραστούν οι ίδιοι νέοι για την κατάστασή του. Θελήσαμε επίση να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των ίδιων των νέων για την κατάσταση των συνομιλικών του σε άλλε χώρε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό ο διασυνοριακό διάλογο δεν λαμβάνει στην πράξη πολύ συχνά χώρα. Είδαμε επίση ότι υπάρχουν διάφορες προκαταλήψεις, διάφορα στερεότυπα, τα οποία υφίστανται ακόμα, το ότι οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ αυστηροί και αδέκαστοι, το ότι οι Έλληνες είναι τεμπέλητες για παράδειγμα. Θεωρήσαμε λοιπόν θα πρέπει να καταρρύψουμε όλα αυτά τα στερεότυπα και να καταφέρουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων εν έτη 2014. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντω υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν υπάρχει ε, ε, ελεύθερη πρόσβαση των νέων στην πολιτική. Θελήσαμε να καταλάβουμε λοιπόν για ποιο λόγο υπάρχουν προβλήματα, για ποιο λόγο πάρα πολλοί νέοι αισθάνονται αποκομμένοι από την πολιτική. Θεωρήσαμε επίση ότι θα έπρεπε να συσπηρωθούμε όλο και περισσότερο εμεί οι νέοι, να μην αισθανόμαστε μονομένοι ο καθένα στη χώρα του, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν ε, σημαντικά προβλήματα, σημαντικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν όλους, ζητήματα τα οποία δεν είναι απλώς εθνικά, αλλά διεθνικά, πανευρωπαϊκά. Θέλησαμε λοιπόν από κοινού να περιγράψουμε το μέλλον το οποίο επιθυμούμε. Θα ήθελα λοιπόν να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα από το διπορικό μας αυτό, βλέπουμε ότι κάθε γενιά αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της. Η δική μας η γενιά έχει τεράστιες προκλήσεις, τόσο προσωπικές όσο και διαρθρωτικές βλέπουμε ότι ε, εμείς χρειαζόμαστε πλέον ένα όραμα, χρειαζόμαστε ελπίδα, χρειαζόμαστε αυτοπεποίθηση και θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό βιώσιμο μέλλον. Πολύ συχνά όμως φοβόμαστε να δημιουργήσουμε οικογένειες, ανησυχούμε πάρα πολύ για την υπερθέρμανση του πλανήτη, για την κλιματική αλλαγή, για την ανεργία, για την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, για τις ε, ανεξέλεγκτες ιδιωτικοποιήσεις Θεωρώ όμω ότι αυτέ είναι οι προκλήσει οι οποίες ναι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε, δεν μπορούμε να απομονωθούμε στην Ευρώπη και να παριστάνουμε ότι τίποτα δεν συμβαίνει από όλα αυτά, ότι τα προβλήματα δεν υφίστανται. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και πρέπει να αναλάβουμε δράση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα όπω η κλιματική αλλαγή, η ανεργία, οι προκλήσει που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το καθεξής. Είμαστε μια γενιά η οποία ενηλικιώνεται σε μια ήπειρο που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν αρκεί για εσάς ή για το σύστημα να μας προσφέρετε απλώς μία απλή λύση. Θεωρούμε ότι η λύση θα πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστική. Πάρα πολλοί νέοι μας είπαν ότι δεν αναζητούμε απλώς μια δουλειά, θέλουμε διαρθρωτικές, σημαντικές, ουσιαστικές αλλαγές στις κοινωνίες μας. Ας είμαστε λοιπόν δημιουργικοί, ας προσπαθήσουμε πραγματικά να αποκριθούμε στις ανάγκες αυτές των νέων, ας τολμήσουμε να πιστέψουμε ότι όντως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν γιατί καταλαβαίνετε ότι προφανώ κάτι δεν πάει καλά όταν η οικονομία δεν είναι σε θέση να προσφέρει ευκαιρίε στου νέου και κάτι δεν πάει καλά όταν το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αποκριθεί και δεν μπορεί να τηθασεύσει ένα ανεξέλεκτο οικονομικό σύστημα το οποίο ενδιαφέρεται μόνο για τον πλουτισμό ορισμένων και δημιουργεί κρίση για όλου του υπόλοιπου. Δεν μπορεί το μέλλον μα να αποφασίσετε από τα χρηματιστήρια, από τι πολυεθνικέ επιχειρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τα συμφέροντα των ίδιων των πολιτών και όχι τα μονομένα συμφέροντα κάποιων πολυεθνικών. Αυτά είναι τα συμπεράσματα ορισμένων λοιπόν νέων οι οποίοι συζήτησαν μαζί μας και ουσιαστικά αυτά είναι και τα αιτήματα τα οποία προωθούν προς εσάς τους πολιτικούς. Να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς κοινωνία και οικονομία και βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι ο καπιταλισμός ανθεί. Αυτό είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι αποφάσισαν να καταλήψουν την Ήπεθρο να πάνε στις πόλεις προκειμένου να γίνουν ε, διευθυντές επιχειρήσεων, designers και το καθεξής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ας μην εκμεταλλευόμαστε τον κόσμο μόνο για το δικό μας προσωπικό οικονομικό συμφέρον, αλλά ας καταφέρουμε να αρχίσουμε να, δράσουμε, να δρούμε διαφορετικά, με έναν τρόπο συλλογικό, με έναν τρόπο υπεύθυνο και συλλογικό, βιώσιμο. Ας μην έχουμε πλέον παροπίδες, Ας καταφέρουμε να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Είδαμε ότι ακριβώς αυτό θέλουν οι Κινέοι της σημερινής εποχής και ελπίζουμε ότι τελικά από την κρίση αυτή την οποία προκάλεσε το κέρδος, η απληστία, θα καταφέρουμε τελικά να αλλάξουμε νοοτροπία. Θα καταφέρουμε να δούμε μια συμπεριφορά όλο και πιο υπεύθυνη, όλο και πιο κοινωνική. Γνωρίζουμε ακριβώς που είναι τα κακό κείμενα, γνωρίζουμε ποιες λύσεις πρέπει να επιφέρουμε. Επιστρέψαμε πάντως στη Δανία ελπίζοντα ότι όντω τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Συντοποιούμε ότι ενδεχομένω η δική μα γενιά να είναι η πρώτη γενιά νέων που θα μπορούσε πραγματικά να επιφέρει την αλλαγή, που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πραγματική ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Έχουμε νέα μέσα στη διάθεσή μα, μπορούμε πλέον και μιλάμε οι περισσότεροι εύκολα αγγλικά, μπορούμε να ταξιδεύουμε σε διάφορε χώρε και πραγματικά να μιλάμε απευθείας με τους ανθρώπους. Επίσης έχουμε στα χέρια μας το διαδίκτυο το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία μας με οποιονδήποτε στην Ευρώπη, ανα πάσα στιγμή. Και έπειτα έχουμε και τα ανοιχτά αυτά σύνορα τα οποία μας επιτρέπουν να ταξιδεύουμε πάρα πολύ εύκολα και να συναντούμε όποιον επιθυμούμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι ενδεχομένω να είναι η δική μας η γενιά που έχει την ευκαιρία να είναι μια πραγματικά αυθεντική ευρωπαϊκή γενιά. Έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μόνο σημείο αφορά στην προηγούμενη γενιά ή τους γονείς μας, πως αυτοί χρησιμοποίησαν δηλαδή τα μέσα τα οποία εμείς έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Επίσης, νομίζουμε ότι στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι να κινητοποιήσει όλη αυτή την πολιτική ενέργεια που υπάρχει στους νέους αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες. Πραγματικά υφίσταται η βούληση αυτή, υφίσταται η ενέργεια αυτή το ένα τρίτο περίπου των ανθρώπων που συναντήσαμε ήδη συμμετέχουν ε, στις ε, εκλογές, είναι σε ηλικία κατά την οποία μπορούν να ψηφίσουν. Δικός μας στόχος, δικό μας καθήκον θα πρέπει να είναι να ξεφύγουμε από τις εθνικές, πολιτικές, κοινωνικές κατηγορίες και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, θα καταφέρουμε να έχουμε όλοι ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον αν από κοινού αναλάβουμε δράση, αν από κοινού διασυνοριακά αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Το πρόγραμμά μα ονομάζεται Our Europe, η Ευρώπη μα για δύο λόγου. Πρώτον, διότι θα πρέπει να αναλάβουμε από κοινού ευθύνη για την ήπειρό μα. δεν μπορούμε να μείνουμε εκτό παιχνιδιού, βρισκόμαστε ήδη μέσα στο παιχνίδι αυτό και πρέπει και εμεί να συμβάλλουμε και κατά δεύτερο λόγο θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει απλώς να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας ή να ζήσουμε ουσιαστικά τα όνειρα ή τα σχέδια άλλων ανθρώπων. Έχουμε και εμείς το δικαίωμα να έχουμε τα δικά μας όνειρα, τις δικές μας απαιτήσει, τις δικές μας προσδοκίες και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δείξουμε το απαραίτητο θάρρος και να πούμε ότι η Ευρώπη αυτή είναι και δική μας Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για το project. Ε, το δεύτερο βραβείο τώρα, Iris Bass και Von Helda. Ε, good afternoon. Ε, Καλησπέρα. Είμαστε μέλη του Γιάου Delft που είναι ένα συμβούλιο νέων στην πόλη του Delft στην Ολλανδία. Είναι ε, νέοι 15 με 22 ετών. Έχουμε 6 ενεργά μέλη και 8 εσωτερικά Προσπαθούμε να οργανώσουμε δραστηριότητες στο Delft και κοντά στο Delft, ιδιαίτερα σχετικά με προβλήματα στον Δήμο, για να έχουμε τη, τη γνώμη των νέων και έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η φωνή των νέων στο Delft για τον Δήμο. Αυτή τη φορά όμως δεν περιοριζόμαστε στον Δήμο του Ντέλφτα αλλά θελήσαμε να δούμε τα πράγματα πανευρωπαϊκά, να εξετάσουμε δηλαδή τη μακροχρόνια ανεργία των νέων. Κάναμε μερικές έρευνες για την ανεργία των νέων στην Ευρώπη και η αριθμή αυτή είναι από το 12. Βλέπετε ότι πρέπει να το προσέξουμε το πρόβλημα γιατί είναι συνεχώς αυξανόμενο. Η παιδεία έχει μεγάλο ρόλο σε αυτό, διότι δίνονται όλο και λιγότερα κονδύλια για σχολεία και πανεπιστήμια. Είναι όλο και πιο δύσκολο για τους φοιτητές να πάρουν δάνεια και να αναλάβουν προγράμματα και χρειάζεται να δουλεύουν εκτός από τις σπουδέ τους για να τις πληρώνουν. Κατά το συνέδριό όμως βασιστήκαμε σε έξι διαφορετικά θέματα. Η κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, γιατί βρήκαμε ότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με εκείνους που θέλουν να εργαστούν εκτός από τη χώρα τους ούτε καν γνωρίζουν ότι μπορούν να το πράξουν μετά η συνεννόηση επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πολλές εταιρείες δεν γνωρίζουν επίσης την κατάσταση των νέων ούτε οι νέοι γνωρίζουν ποιες εταιρείε θα ήθελαν να αναλάβουν προγράμματα με φοιτητέ. Μετά η αναγνώριση των διπλωμάτων, όπου είδαμε ότι δεν θεωρούνται ισότιμα όλα τα διπλώματα στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος σύγκρισης που δεν υπάρχει πανενουσιακός. Οι νέοι επιχειρηματίες και το επιχειρηματικό πνεύμα Πολλοί νέοι θέλουν να αρχίσουν μια επιχείρηση, αλλά δεν υπάρχουν επίσης οδηγίες και πληροφορίες για αυτούς. Οι σπουδές χωρίς σύνορα είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό, όπως το πρόγραμμα Έρασμος που είναι κάτι πολύ θετικό, αλλά δεν επωφελούνται όλοι οι φοιτητές από τέτοια προγράμματα και το τελευταίο σημείο που συζητήσαμε ήταν οι υποτροφίες ή μάλλον οι μαθητείες γιατί μπορεί πολλοί να τις θεωρήσουν σαν απλώς φτηνή εργασία για τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό κάναμε και ένα ψήφισμα περί αυτού. Τα ερωτήματά μας τα στείλαμε τα δείξαμε, τα συζητήσαμε με όλους όσους συμμετέσχουν στο συνέδριο. Στην αρχή όλοι μαζί και μετά αναομάδες για να έχουμε ορισμένα συμπεράσματα πριν να γίνει το ψήφισμα. ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει πράγματι τη συζήτηση που είχε γίνει σε διεθνή κλίμακα. Τα θέσαμε μερικά ερωτήματα αλλά και σε τοπική γιατί δεν είναι σημαντικό μόνο να συζητούμε για ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και τι μπορεί να γίνει και τοπικά. Μπορεί κανείς να αρχίσει σε μικρή κλίμακα και μετά να αυξηθεί η δραστηριότητα αλλά ως άτομο δεν μπορεί να κάνει πολλά. Πανενουσιακός μπορεί όμως να κάνει πολλά τοπικός. Τον Νοέμβριο του 12 λοιπόν καλέσαμε 60 νέους από 10 διαφορετικές χώρες στο Ντέλφτ για να συζητήσουμε αυτά που σας είπαμε. Μίλησαν πολλοί από αυτούς, ας πούμε κάποιος από την οργάνωσή μας και κάναμε και ορισμένα brainstorming δύο την ημέρα και τελικά έβγαινε ψήφισμα όσων θεμάτων είχαμε συζητήσει. Στο τέλος της εβδομάδας όλα αυτά τα ψηφίσματα συνθέσαμε σε ένα με κάποιες ψηφοφορίες. Βάλαμε στον τοίχο αφήσει με όλα τα ψηφίσματα και οι νέοι μπορούσαν έτσι να δουν τι ήθελαν να αλλάξει ή τι θεωρούσαν σημαντικότερο. Να πώς περνούσαμε την ημέρα μας. Στην αρχή γινόταν μια περίληψη των δραστηριοτήτων της ημέρας, μετά τον πρώτο brainstorm, μετά ένα μίνι ψήφισμα μετά το γεύμα και μετά το δεύτερο brainstorm και γραφόταν το δεύτερο μήνυ ψήφισμα. Και τελικά συζητιούνταν όλα τα θέματα που συζητήθηκαν σήμερα. Στο βραδινό πρόγραμμα περάσαμε πολύ καλά και για να γνωριστούμε καλύτερα γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν και αυτό σημαντικό να γνωριζόμαστε καλά ως ομάδες γιατί έτσι ελπίζαμε ότι ο καθένας θα ανοιγόταν περισσότερο και θα μιλούσε πιο εύκολα για τα προβλήματά του. Στο τέλος της εβδομάδας, όπως σας είπα, κάναμε ένα γενικό ψήφισμα για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Πρώτον για τις μαθητιές. Αυτό μπορεί να ωφελήσει την Ένωση γιατί ε, δίνει πληροφορίες στον νέο για την πραγματική εργασία που μπορεί να κάνει να παίξει το ρόλο όχι μόνο του υπαλλήλου αλλά καμιά φορά και του εργοδότη. Η εμπειρία της εργασίας σε πολλές επιχειρήσεις δεν ήταν μόνο θετική όμως πρέπει να προωθηθεί η σημασία που έχουν οι μαθητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης νομίζουμε ότι το επιχειρησιακό επιχειρηματικό πνεύμα των νέων είναι επίσης σημαντικό και πρέπει να στηριχθεί γιατί μπορεί έτσι να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων, να δημιουργηθεί θέσεις απασχόληση και γενικότερα να βοηθηθεί η οικονομία της Ένωσης σε τρία επίπεδα. Πρώτον, να τα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτικά ή με κάποιον άλλο τρόπο. Δεύτερον, συστήνουμε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στα σχολεία για να διευκολύνονται οι δυνατότητες των νέων για μαθητεία και για να μπορούν να αρχίσουν την επιχείρησή τους. Και τέλος, θα ήταν θετικό και για τις υπάρχουσες μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις αν βοηθήσουν τους νέους να επιχειρήσουν. Και για την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας θεωρούμε σημαντικό να αυξηθεί η πληροφόρηση που υπάρχει για τις δυνατότητες εργασίας σε τρίτη χώρα. Γιατί οι Έλληνες, οι νέοι δεν τα γνωρίζουν αυτά, δεν έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Επίσης θα θέλαμε να είναι η πληροφόρηση αυτή και σωστή και εύληπτη ώστε να μπορεί κανείς να πάει κάπου αλλού να εργαστεί. Για την ισοτιμία των διπλωμάτων τώρα θα θέλαμε να υπάρχουν συγκρίσιμα προσόντα για τα διάφορα μαθήματα ώστε να μπορεί κανείς αμέσως να δει σε τι επίπεδο βρίσκεται συγκρίσιμα με άλλων σχολών ή πανεπιστημίων για να το γνωρίζουν αυτό και οι εργοδότες. και να μπορέσουν και τα πανεπιστήμια αν χρειαστεί να αυξήσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουν και τα διπλώματά τους. Όσο για τη λεγόμενη cross-fertilization, Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό. Επίσης, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ο ένας την προοπτική του άλλου και όλα αυτά να είναι πιο προσβάσιμα ώστε να καταλήξουν σε καλύτερη αμοιβαία πληροφόρηση ή cross-fertilization που λέμε. Έχουμε λοιπόν σχέδια όχι μόνο για την Ένωση, αλλά και τοπικά. Και επειδή ήρθαν νέοι στο Τέλφτα από διάφορες χώρες, Θέλησαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει και στην πόλη μας, στο Delft. Δύο προγράμματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το πρώτο λέγεται Werken in Delft που είναι μια σελίδα facebook όπου μπορεί κανείς να ανεβάζει μικρές αγγελίες για δουλειές και έτσι ελπίζουμε να είναι ευκολότερο για τους νέους αυτούς να ψάξουν για δουλειά και να βρουν. Και έχουμε και ένα pop-up store όπου νέοι που δεν ξέρουν πώς να αρχίσουν την επιχείρησή τους ή πώς να γράφουν το βιογραφικό τους. Μπορούν να πάνε σε αυτό το pop-up store όπου θα, άλλοι νέοι θα τους πληροφορήσουν για να μάθουν καλύτερα πώς βρίσκουν δουλειά και πώς γράφουν βιογραφικά κλπ. Εδώ βλέπετε μία φωτογραφία των 50 νέων που συμμετέσχουν στο συνέδριό μας και νέα πολιτικούς από διάφορες άλλες πόλεις έξω από τον Τέλφτ πριν από δύο χρόνια. Ε, από τότε έχουν γίνει πολλά αλλά δεν έχουν τελειώσει. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας κατά της ανεργίας των νέων ώστε να έχουν κάποιο μέλλον. Σας κατευχαριστώ. Thank you, Σε ευχαριστώ, Η επόμενη, η τρίτη νικητές, η Χριστιανά και η Ευανθία. Hi, we Γεια σας, είμαστε η Χριστιανά και η Εύα από την Κύπρο. Είμαστε μέλη της άτυπης ομάδας Youth Dynamics και είμαστε εθελοντές, η ομάδα εθελοντών από την Κύπρο και η ομάδα μας δημιουργήθηκε το 2011 μετά από ανταλλαγές απόψεων και προγράμματα που είχαμε στο εξωτερικό, θερήσαμε την εμπειρία αυτή να τη μεταφέρουμε και στη δική μας κοινότητα. Το σχέδιο όμως λοιπόν, το project μας ήταν Employment for You, μία κατάρτιση για τους νέους. Σε αυτό συμμετείχαν το πρόγραμμα εννέα χώρες, η Κύπρος, η Εστονία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετωνία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Ισπανία. Είχαμε σύνολο 26 συμμετεχόντων στο σχέδιο αυτό, στο project αυτό. Οι περισσότεροι από τους νέους που συμμετείχαν ήταν άνεργοι και νέοι που έψαχναν μια θέση απασχόλησης τότε. Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στην Ευκοσία και Οργανώσαμε αυτό το project 13 με 20 Απριλίου του 2013. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Λευκοσία μπόρεσαν οι συμμετέχοντες να επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς μας χώρους και να μάθουν για την ιστορία της Κύπρου. Πού έλαβε χώρα το project αυτό. Στον ε, ξενώνα νέα της Λευκοσίας Πριν αρχίσουμε την κατάρτιση, δείξαμε στους ε, συμμετέχοντες πώς ήταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Κύπρο και στις περισσότερες χώρες οι οποίες αντιμετώπιζαν ε, μια οικονομική κρίση. Και είδαμε ποια ήταν η διαδρομή, τελειώνει ε, κανείς ε, ποια είναι η διαδρομή που ακολουθεί κανείς. Τελειώσει στο σχολείο, κάνει σπουδές, ε, εργάζεται και στο τέλος παίρνει σύνταξη. Αυτό για τους προηγούμενους. Σήμερα τα πράγματα είναι τελώ διαφορετικά. Τελειώνουν ε, τα παιδιά το σχολείο, έχουν περιόδους μαθητείας, μπορούν να φύγουν, να κάνουν μια άλλη εξειδίκευση, να πάρουν ένα πιστοποιητικό ή το πτυχίο τους, να ακολουθήσουν άλλες ε, σπουδές, άλλη εξειδίκευση και όπως είδαμε το ποσοστό ενεργείας στην Ευρώπη και κυρίως στις χώρες αυτές είναι Τους είπαμε πώς μπορεί κανείς να ψάξει, να βρει ε, δουλειά, πώς ε, μπορεί να, ποια διαδικασία ακολουθήσει, ποιε είναι οι ξενοτόμες δεξιότητες, πώς μπορεί κανείς με δημιουργικότητα και με πνεύμα επιχειρηματικότητας να πετύχει και ποιος είναι ο ρόλος των οργανώσεων νέων, των κυβερνήσεων, των συμβουλίων νέων και των οργανώσεων. Και βεβαίως ποιες είναι οι δυνατότητες όταν τελειώσει το σχολείο, τι μπορούν να κάνουν. Κάτι άλλο που τους αποδείξαμε ήταν να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι εάν φτάσει κανείς λίγο πριν από το διέξοδο, πάντα μπορεί να προχωρήσει και να είναι δημιουργικός, διότι ξέρουμε ότι πολλούς νέους τους απασχολεί η ενεργεία, πολλοί έχουν και κατάθλιψη και πρέπει κάτι να κάνουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Μία από τις δραστηριότητε που είχαμε την ονομάσαμε Καφενείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες συμμετέχοντες, έκαναν ερωτήσεις, απαντούσαν του τύπου τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης για να προωθήσουν την θέση απασχόλησης, οι νέοι, οι οργανώσεις των νέων, οι εργαζόμενοι. Έγιναν λοιπόν συζητήσεις μεταξύ των μελών της ομάδος και παρουσίαζε κάθε ομάδα στην άλλη τα αποτελέσματα στο οποίο κατέληξε. Επίσης υπήρχε ένα εργαστήριο για το ε, Europass CV, για το περίφημο αυτό ευρωπαϊκό ε, βιογραφικό που πρέπει να έχει κανείς και πώς το συμπληρώνει. Και πώς ε, παρουσιάζεται κανείς όταν έχει συνέντευξη για να ζητήσει συνεργασία, Πώς δίνει το χέρι, κάνει τη χειραψία, πώς πρέπει να είναι ντυμένος, πρέπει να ε, συμπεριφερθεί για να κάνει καλή εντύπωση στον μελλοντικό εργοδότη ενδεχομένω. Uh, e Επίσης έγινε μια παρουσίαση για την ε, επαγγελματική σταδιοδρομία, της καριέρας επαγγελματικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σταδιακά τους δείξαμε πώς μπορεί κανείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει αίτηση για μια θέση απασχόλησης. Επόμενο εργαστήριο με τους νέους, σχέδιο ε, Inspire και Lead, ε, έμπνευση και τρόπος με τον οποίο θα ηγηθείς ένα τέτοιο σχέδιο. Δεν να λες κανένα νέο να του κάνει κανείς μάθημα εξ κάτεντρα. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς με δημιουργικό τρόπο να πείσει τους νέους να κάνουν το δικό τους σχέδιο για να το εφαρμόσουν ε, όταν θα φτάσουν στη χώρα τους. Και πολλοί μας είπαν ότι ε, χρησιμοποιούσαν τα διάφορα προγράμματα τα οποία μάθαν, θα τα μετέφεραν στις χώρες τους, στις οργανώσεις νέων για να τα χρησιμοποιήσουν σωστά και να επωφεληθούν από την εμπειρία. Επίσης, μια άλλη παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ε, Κύπρο. Εξηγήθηκε τώρα το οποίο δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι περισσότεροι νέοι δεν ήξεραν περί τίνος πρόκειται. Δεν ήξεραν πώς ε, ε, λειτουργούν οι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η επόμενη παρουσίαση που κάναμε έγινε από κάποιον άλλο αξιωματούχο, ο οποίος τους μίλησε για οικονομικά προβλήματα, για τη χρηματοπιστωτική κρίση και είπαμε ότι ο καθένας θα πρέπει να επισημάνει τα προβλήματα τα σχετικά τα οικονομικά στη χώρα του. Επίσης, μια άλλη παρουσίαση εκ μέρους ε, της υπηρεσίας ε, που ασχολείται με θέματα ανθρωπίνου δυναμικού στην Κύπρο. Πώς μπορεί να ψάξει κανείς να βρει δουλειά σε δύσκολες ε, συνθήκες εργασίας ε, στην αγορά σήμερα, πώς μπορούν να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα, ποιε είναι τα προσόντα και οι δεξιότητες που χρειάζονται, πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Επίσης είχαμε μια άλλη παρουσίαση για τα προγράμματα ε, η νεολαία σε δράση, ποιες είναι οι δράσεις κλειδιά και μία νέα κοπέλα από την Κύπρο μας είπε ποια ήταν η προσωπική της εμπειρία και πώς υποβελήθηκε από το ότι συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα μαθητείας στην Ευρώπη για έξι μήνες και μετά πώς ό,τι έμαθε μπόρεσε να το εφαρμόσει ε, και εργάστηκε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ε, της προσφοράς εθελοντικής εργασίας μεταξύ των νέων. Επίσης, ε, μιλήσαμε για το πώς μπορεί ο καθένας να λειτουργήσει μέσα σε μία μικρή, μία, ευρω... κυβερνητική οργάνωση, την οποία επίση μπορεί να συστήσει ο ίδιος, και ε, εμπλουτιστήκαμε από τις εμπειρίες και την κουλτούρα και τις ανταλλαγές απόψεων όλων. Ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος στο τέλος κάθε ημέρας να έχουμε και μία μικρή παρουσίαση από κάθε χώρα για τις παραδόσεις και τα πολιτιστικά κάθε χρόνος. Κάναμε επίσης και ένα ταξίδι στην Μεσό, εδώ βλέπετε τις φωτογραφίες. Και ήταν εξαιρετικό το ταξίδι αυτό, ένα ταξίδι επιτόπου όταν είστε κάπου είναι πολύ καλό διότι μπορεί ε, ε, να δει με τα ίδια του τα μάτια πώς έχει η παράδοση και η κουλτούρα κάθε χώρα. Εμείς προσπαθήσαμε να τους δείξουμε ό,τι μπορούσαμε, ξέρουμε ότι η Κύπρος είναι μακριά από την υπόλοιπη Ευρώπη και κλείσαμε με τα μελλοντικά σχέδια. Θέλουμε, ε, είμαστε ε, εθελοντές, είμαστε καθηγητές, θα θέλαμε αυτή η άτυπη ομάδα να... Ε, αναπτυχθεί περισσότερο, να συνεχίσει τις δραστηριότητες για να δει αν μπορεί να λύσει προβλήματα όπως αυτό της ανεργίας. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες συμμετοχές από νέους σε εθνικό και διεθνές ε, επίπεδο. Θα θέλαμε να εμπνεύσουμε τους άλλους, να δημιουργήσουμε κύρνητρα, να ενημερώσουμε με δημιουργικότητα για να ενισχυθεί η θέση τους. Και νομίζω ότι με την ε, η εκπαίδευση ε, έχει και άμεση σχέση με την ε, ανεργία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία τελειώνουν το σχολείο και εξαιτία του περιβάλλοντό τους δεν ξέρουν τι να κάνουν ίσως, κατευθύνονται στο πανεπιστήμιο, παίρνουν ένα πτυχίο και μετά δεν ξέρουν τι να το κάνουν το πτυχίο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν και στην παιδεία κάτι να αλλάξει, να υπάρχει περισσότερη δημιουργικότητα, δημιουργικότητα η οποία λείπει και από τα σχολικές αίθουσες και πολλές φορές οι καθηγητές οι ίδιοι δεν εμπνέουν τα νέα παιδιά, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και η παιδεία νομίζω ότι αν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό θα βοηθήσει να λύσουμε και ένα μεγάλο μέρος της ανεργίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ωραία και ενδιαφέρουσα, τις ωραίες και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο τώρα για να κάνετε ερωτήσεις, να κάνετε σχόλια μετά από τις παρουσιάσεις των νέων παιδιών. Ε, Mrs. Κυρία Κάμερβερτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και συγχαίρω τις τρεις ομάδες των νικητών. Εδώ και πέντε χρόνια είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Γερμανικής Επιτροπής που απονέμει το βραβείο Καρλομάγνου και κάθε φορά με εκπλήσει η δημιουργικότητα και η δέσμευση των ε, νέων και είδαμε πόσο ενδιαφέροντα είναι τα προγράμματα που μας παρουσιάστηκαν. Πάντα εκπλήσαμε λοιπόν θετικά. Εάν μπορούσαν τα σχέδιά σας να είναι ε, αντιπροσωπευτικά της ε, νεολαίας μας στην Ευρώπη, δεν θα είχαμε να φοβηθούμε τίποτε για τους νέους και θα πρέπει όλοι να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Βεβαίως, εάν όλοι οι νέοι ε, σκέφτονταν όπως και εσείς και αν σκέφτονταν τα ίδια πράγματα την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε ήσυχοι. Δεν έχουν όμως έτσι τα πράγματα. Ξέρουμε ότι εσείς είστε μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Ένα ερώτημα προς τους νικητές. Ξέρω ότι κάνατε αρκετά ταξίδια, αλλά και άλλοι δικαιούχοι των ε, προγραμμάτων εποφελήθηκαν τι είδατε εσείς ταξιδεύοντας και μιλώντας με τους άλλους. Υπάρχει ίδια αντίληψη ε, μεταξύ όλων για τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχει μια ενιαία άποψη ή διαπιστώσατε ότι ανάλογα με το κράτος μέλος το οποίο ανήκει κανένας υπάρχουν μεγάλες ε, ε, διαφορές. Κυρίως σκέφτομαι τις χώρες οι οποίες μας στείλουν από την οικονομική κρίση είναι πιο αρνητικοί οι νέοι εκεί όσον αφορά τον μέλλον τους ή Κυρίως αντιθέτως στις χώρες αυτές υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία και θέλουν οι νέοι να κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεπεράσουν τον οικονομικό μαρασμό των χωρών τους. Äh, Ποιε είναι επί του θέματος η δική σας άποψη, ποια είναι η εμπειρία σας. Με ενδιαφέρει να την ακούσω. Επίσης, τα προγράμματά σας συνεισέφεραν κατά τον α ή β λόγο ώστε να αποτελέσουν έναυσμα για νέους ε, να πάρουν την κατάσταση για το μέλλον στα χέρια τους αντί να κάνουν επικρίσεις επί επικρίσεων. Κυρίως τους ε, δανούς απευθύνομαι, διότι από ό,τι κατάλαβα θέλετε να κάνετε τους νέους πιο ανεξάρτητους ώστε να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον τους. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση των προγραμμάτων, των σχεδίσεων και ελπίζω ότι αυτό που κάνετε θα έχει μία διάρκεια στο χρόνο και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και την εξέλιξη των προγραμμάτων που θέσετε σε εφαρμογή. Ευχαριστώ. Time, so uh, I have λείπει ο χρόνος. Να κλείσω τον κατάλογο των μιλητών. Εντάξει μετά τον κύριο Γραμματικά και κλείνει. Κυρία Φερχάιν. θα αρχίσω ευχαριστώντας σας όλους πολύ θερμά. Είναι μεγάλο κατόρθωμα νομίζω αυτά που ακούσαμε σήμερα διότι τα project όλα αυτά για το βραβείο Καρλομάγνου μου άρεσαν πολύ. Έχω πάει και εγώ ως μέλος επιλεκτικής ομάδας σε διάφορους διαγωνισμούς. Ήμουν και δήμαρχος του Άχεν και έχω συναντήσει και στην οι υποψηφίους. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ ωραίο που μπορέσατε σήμερα να έρθετε να μας παρουσιάσετε τα σχέδιά σας. Γιατί έτσι βλέπουμε ότι έχουν πολλά μας πούν οι νέοι που ασχολούνται με το μέλλον τους και συναντούν και άλλους νέους και βλέπουν ποιες ανάγκες έχουν για να συνεννοηθούν όχι παθητικά μόνο ή απαθητικά να, αλλά με ενεργό τρόπο δημιουργώντας δικά τους σχέδια και προγράμματα και projects και συζητώντας τα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που ήρθατε να μας τα πείτε. Τώρα αναρωτιέμαι κατά πόσον είναι βιώσιμα αυτά τα προγράμματα ή τέτοια προγράμματα και πώς θα μπορούσαν κι άλλοι νέοι να συμμετάσχουν σε ανάλογα. Ε, σας ρωτάω λοιπόν, έχετε καμία πρόταση για μας τι μπορούμε να κάνουμε ως ευρωβουλευτές δηλαδή για να βελτιώσουμε τα πράγματα ώστε να μπορούμε να κάνουμε τους νέους να αισθάνονται πιο κοντά στην Ευρώπη γιατί καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι ενώ έρχονται πολλοί επισκέπτες και ολόκληρα σχολεία καμιά φορά στις Βρυξέλλες ε, δεν έχουν όλοι το ίδιο ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Πολλά εξαρτώνται από το κατά πόσον ο δάσκαλος που του συνοδεύει ενδιαφέρεται. Αλλά βέβαια υπάρχει και η προσωπική, το προσωπικό ενδιαφέρον των νέων και των μαθητών και φοιτητών. Αν ενδιαφέρονται δηλαδή για τίποτε παραπέρα από το άμεσο περιβάλλον τους. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε τίποτε παραπάνω για να φτάσουμε στους νέους, να τους πληροφορήσουμε περισσότερο για τα ευρωπαϊκά, την ευρωπαϊκή πολιτική και να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Ίσως καμιά φορά ακούνε πάρα πολλά οι νέοι, πάρα πολλά μηνύματα και συγχέονται. Είναι δύσκολο βέβαια να, να ενθουσιάσουμε τους νέους για την Ευρώπη. Εσείς μάλλον ήσασταν ήδη ανοιχτοί ως νοοτροπία στο ευρωπαϊκό, στον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Ερωτώ λοιπόν για τέταρτη φορά πώς νομίζετε ότι μπορούμε να πείσουμε τους νέους να γίνουν πιο ενθουσιώδεις περί αυτής. Ευχαριστώ κυρία Βόρτ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Και εγώ συμμετέχω σε τέτοια προγράμματα και πραγματικά ενθαρρύνω τους νέους να ταξιδεύουν και να μοιράζονται αυτές τις διαφορετικές απόψεις διασυνοριακά. Πραγματικά λοιπόν να σας συγχαίρω για τα όσα έχετε κάνει. Νομίζω ότι η φιλοδοξία σας είναι όντω πολύ μεγάλη και θα πρέπει να τη χαιρετήσουμε. Μ' άρεσε ιδιαίτερα το ότι η δεύτερη ομάδα, μάλλον η ομάδα από την Κύπρο μας είπε πόσο σημαντική είναι η δημιουργικότητα, ότι είναι πολύ δύσκολο κανείς να καταφέρει να αξιολογήσει το βαθμό δημιουργικότητας στα πλαίσια ενός στήρου βιογραφικού, ενώ όλοι συνειδητοποιούμε ότι η δημιουργικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ποιε είναι οι χώρε που δεν επισκεφθήκατε, ρωτώ του Δανού αυτή τη στιγμή, γιατί είπατε ότι πήγατε σε 24 ευρωπαϊκέ χώρε. Ποιε είναι οι τρει χώρε που δεν επισκεφθήκατε, και μάλιστα το project σα έγινε πρωτού ενταχθεί η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι. Εγώ εκπροσωπώ εδώ τη Μεγάλη Βρετανία, τα αγγλικά είναι η μητρική μου γλώσσα και μου έκανε εντύπωση που είπατε ότι χρησιμοποίησατε τελικά την αγγλική γλώσσα προκειμένου να συνεννοηθείτε με άλλους νέους. Και θα θέλω ουσιαστικά αυτό να το χρησιμοποιήσω και σαν θετικό επιχείρημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική μου τη χώρα. Όπως ξέρετε υπάρχουν ε, σημαντικές ανησυχητικές αργατάσεις ευρωσκεπτικισμού. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να πούμε και στους ίδιους τους Άγγλους ότι η αγγλική γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να φέρει κοντά τους νέους. Είναι ουσιαστική σημασία η αγγλική γλώσσα, όπως είπατε και εσείς, για τα δικά σας τα προγράμματα. Θεωρώ λοιπόν ότι χρησιμοποιώντας το επιχείρημα αυτό θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε περισσότερο και τους νέους στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να διαφερθούν και τα δικά σας τα προγράμματα. Δεν ξέρω αν έχετε τις σελίδες Facebook ή Twitter γιατί θα ήταν πιστεύω ενδιαφέρον και στις παρουσιάσεις σας να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι διευθύνσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο Facebook ή στο Twitter για να συνδεθούμε μαζί σας. Σας ε, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχετε δύο λεπτά στο τέλος για να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Η κυρία Σρέντεβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα σας μιλήσω γαλλικά. Ίσως να με καταλαβαίνετε καλύτερα από ότι αν μιλούσα τσέχικα που είναι η μητρική μου γλώσσα. Ήμουν και εγώ μέλος ε, επιλεκτικής ομάδας Εξεταστικής Επιτροπής και μάλιστα συμμετείχα και εγώ στις ε, δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Νέων. Ξέρετε ότι έχουμε μία αντίστοιχη ομάδα και στην ε, Τσεχική Βουλή, η οποία ασχολείται με ζητήματα τα οποία απασχόλησαν και εσά. Πρέπει να σας πω ότι τα συμπεράσματά σας πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για μένα. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι εμείς, οι Ευρωβουλευτές, είμαστε σε θέση μέσω αυτής της ανταλλαγής απόψεων να ενημερωνόμαστε για τις δικές σας εμπειρίες. Σας διαβεβαιώ ότι για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζω πώς σκέφτεστε, ποιες είναι οι απόψεις σας και ποιες είναι οι προτάσεις σα Μία έκκληση θα ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή, θα μπορούσατε στα πλαίσια των project αυτών ή κάποιων μελλοντικών project να επισκεφτείτε και τη χώρα μου, την Τσεχική Δημοκρατία και απευθυνόμενοι στους νέους από την Κύπρο θα ήθελα να σας πω ότι ε, η Τσεχική Δημοκρατία έχει κάποιες πολύ θετικές εμπειρίες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον εκπαιδευτικό τομέα. Ενδεχομένως η εμπειρία λοιπόν της χώρας μου να μπορούσε να σας ενδιέφερε ή να αποτελούσε κίνητρο για αντίστοιχε δραστηριότητες στη δική σας τη χώρα. Σας καλώ λοιπόν να έρθετε στην Τσεχική Δημοκρατία και ενδεχομένως εκεί όντως να καταφέρετε να ακούσετε πράγματα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για σας. Σε κάθε περίπτωση σας καλώ να συνεχίσετε την προσπάθειά σας, σας καλώ να συνεχίσετε να πρεσβεύετε τις ιδέες σας και να συνεχίσετε με τη δραστηριότητα σας αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. And Mr. Uh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς αγαπητοί προσκεκλημένοι για τις παρουσιάσεις σας. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η παρουσίαση των Δανών και των Κυπρίων, όπου αναφέρθηκαν πάρα πολύ σε επιτόπιες δράσεις. Ήρθανε σε επαφή από ό,τι είδα πολλές φορές ακόμα και με ηθήνονται σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά την περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιήθηκαν. Επίσης είπανε τουλάχιστον οι νέοι στα πλαίσια τη παρουσία τη Κύπρου, ότι δεν γνωρίζουν πάρα πολύ νέοι πώ λειτουργούν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν προκειμένου. Επίσης, να αναφερθώ στην παρουσίαση των Δανών. Δεν ξέρω αν κατάλαβα πολύ καλά. Πάντως, σε κάποια στιγμή είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε δημοκρατικό έλεγχο, να τελέσουμε, να ασχοληθούμε με το δημοκρατικό έλεγχο των πολυεθνικών. Αυτό κάπως με ανησυχεί, ακούγεται λίγο περίεργο. Ουσιαστικά αναφέρεστε εδώ πέρα σε μια διαφορετική Ευρώπη, η οποία έπαψε να υπάρχει εδώ και 25 χρόνια. Πάντως, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας, χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τόσες καλές προτάσεις για την ε, συνεργασία επιχειρήσεων και σχολείων, πανεπιστημίων. Σε σχέση με αυτά που είπαν οι προαλήσαντες τώρα, θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι ε, αναφερθήκατε πάρα πολύ συχνά στην αλλαγή. Είπατε ότι πάρα πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει πολύ πιο συγκεκριμένα να μα πείτε ποια αλλαγή θέλετε και ποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν σύμφωνα με εσά. Σας ευχαριστούμε και Γραμματικάκης, έχει το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, πριν γίνω ευρωβουλευτή, ε, ήμουν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και θα ήθελα πάρα πολύ να έχω αυτά τα νέα παιδιά φοιτητέ μου γιατί δείξανε μεγάλη έμπνευση, έκαναν πολύ κόπο, φαντάζομαι τι δυσκολίες αντιμετώπισαν και έτσι θα τους έδινα προκαταρτικά ένα πολύ ωραίο πτυχίο. Σήμερα όμως που η μοίρα το έφερε να είμαι ευρωβουλευτής, δεν θα ήθελα να είναι φοιτητέ μου. Γιατί δεν έχω τίποτα να τους απαντήσω σε όσα είπανε. Και μάλιστα ξέροντας ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά από την Κύπρο ζουν και μια ξενική κατοχή, ότι όλα τα παιδιά της Ευρώπης έχουν αυτή τη φοβερή ανασφάλεια για το μέλλον τους, ότι αγωνίζονται να επιβιώσουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Το μόνο που θα είχα να τους πω σήμερα στα παιδιά όλης της Ευρώπης εκ μέρους όλων μας νομίζω εμάς των μεγαλύτερων είναι μια συγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ομάδα για να απαντήσει. Αρχίζουμε με τους πρώτους νικητές, νικητές του πρώτου βραβείου. Πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η συζήτηση για την πολυεθνικές και για την Σοβιετική Ένωση δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά δεν είμαι με τη μεριά των ε, Σοβιετικών ούτως ή άλλως. Το εξή παράδοξο. Όταν θέλει κανείς να μιλήσει και κίνητα για τις αλλαγές, Είδαμε μεταξύ των προοδευτικών νέων κυρίων στην Νότια Ευρώπη ότι εξαιτία των μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα, κινητικότητα και βούληση να αλλάξουν τα πράγματα. Στις σκανδιναβικές χώρες δεν έχουμε αυτού του είδους τον ενθουσιασμό γιατί σχεδόν τα έχουμε όλα και έχουμε, αλλά έχουμε προβλήματα υπαρξιακά. Άρα δεν έχουμε τα ίδια κίνητρα να μας εμπνέουν. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των, τα, της εμπειρίας μας μετά από το ταξίδι μας στην Ευρώπη. Αν τα νεαρά παιδιά μπορούσαν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε εμείς την κατάθλιψη από τον Νότο, εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τη διαφθορά. Επίσης, σε ερωτήσεις σας, θέσατε το ερώτημα, είμαστε Μπορούμε να ενεργήσουμε δυναμικά ή πρέπει παθητικά να βλέπουμε τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως εξαρτώμεθα από κάποια πράγματα που μας κάνει κάπως παθητικούς, αλλά πρέπει να είμαστε δημιουργητικοί και δυναμικοί. Τώρα είπατε ότι θα πρέπει, θα πρέπει κάποιοι να έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία ευρωπαϊκής κοινωνικοποίησης μάλλον και να μην κλείνεται ο καθένας και να μην περιχαρακώνεται στη χώρα του. Βέβαια, εμείς για περίπου 30 ώρες ε, ασχοληθήκαμε με τα θέματα τα ευρωπαϊκά. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Πώς μπορούμε να ξέρουμε και γιατί ψηφίζουμε στις ε, ευρωεκλογέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη γνώση για την Ευρώπη. Και θα πρέπει κάτι να κάνουμε να αισθανθούμε όλοι περισσότεροι, περισσότερο Ευρωπαίοι. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε όλους τους νέους της Ευρώπης για να τους ενημερώσουμε για το τι είναι η Ευρώπη να τους στείλουμε ταξίδι παντού. Νομίζω όμως θα πρέπει το θέμα κάποιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων να τα δείτε ώστε να περιέχουν περισσότερο την διάσταση Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε αυτό. Εμείς όταν πηγαίνουμε στα διάφορα σχολεία και λέμε στους νέους Ευρωπαίους ποια είναι η εμπειρία μας από την κρίση και στις άλλες χώρες μεταξύ των νέων και στην Ευρώπη τους δείχνουμε φωτογραφίες, βίντεο, και ηχογραφήσεις που έχουμε κάνει στο ταξίδι μας, τι βλέπουμε. Ότι ανοίγεται η Ευρώπη μπροστά στα μάτια των νέων με διαφορετικό τρόπο. Και θέλουν ε, να συμμετάσχουν περισσότερο οι νέοι στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Δεν ξέρουν με ποιο τρόπο. Και μετά μας λένε και οι καθηγητές τους ότι ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η αρχή που κάναμε μιλώντας για το ταξίδι μας και για την Ευρώπη. Και χρησιμοποίησαμε τη δική μας εμπειρία και συγκεκριμένα παραδείγματα από συγκεκριμένες καταστάσεις που αντιμετώπισαν νέοι στην Ευρώπη. Και ως νέοι ίσως δεν έχουμε πάρα πολύ ανεπτυγμένη ακόμη την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα Δέκα δευτερόλεπτα παρακαλώ. Επισκεφθήκαμε 24 χώρες. Δεν επισκεφθήκαμε τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Κύπρο και κάποια άλλη χώρα, αλλά έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ιστότοπο. Ε, μπορείτε να δείτε τι έχουμε κάνει. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρακαλούμε όποια άλλη χώρα θέλει να μας καλέσει. Ευχαριστώ. Η Ολλανδία, για δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τα ευγενικά σας λόγια. Πιστεύω ότι υπάρχουν ανάλογα με την κάθε χώρα και διαφορετικές προοπτικές διότι το γενικό το μισό ότι φοβούν το μέλλον τους είναι και κατά την ε, διάρκεια της επισκευμένης στην Πολωνία μας είπε μια κοπέλα ότι πολλές φορές τα νέα παιδιά τα κυνηγάει η αστυνομία διότι κάνουν διαδήλωση ή δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Αυτό είναι ανησυχητικό. Και η Ευρώπη δεν πρέπει να ανησυχεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να αρχίσουν να συνειδητοποιούν οι νέοι ότι πρέπει να εισακουστεί η φωνή τους. Πολλοί νέοι όμως δεν ξέρουν πώς να το καταρθώσουν αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι τα προγράμματα που μπορεί να οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι θεωρητικά καλά, αλλά τα γνωρίζουν οι νέοι, ξέρουν πώς να συμμετάσχουν. Ούτε καν ξέρουν ότι υπάρχουν τέτοιες προγράμματα. Κάποιος ερώτησε τι λύσεις προτείνεται. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ των νέων, ακόμη και των παιδιών, των νέων που δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Διότι όσοι έχουν πρόσβαση στην ε, ανώτατη εκπαίδευση έχουν και την δυνατότητα να ταξιδεύουν στο, εξωτερικό, στο εξωτερικό, εκτός χώρας τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα και στα άλλα παιδιά. Είναι σημαντικό για να μάθουν καλύτερα την Ευρώπη και να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πραγματική ένωση. Και μπορεί κανείς να πάει σε μια ξένη χώρα και να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ή να βρει δουλειά. Πιστεύουμε επίσης ότι δεν υπάρχει σωστή καθοδήγηση, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση ακόμη και εντός της χώρας του καθενός. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστούμε. Η τρίτη ομάδα. Ένα από τα μέλη μας τα πιο δραστήρια είναι ένα νέο γόρι, το οποίο μας άκουσε μια μέρα να περπατάμε στο δρόμο και να μιλάμε αγγλικά και ήρθε αυθόρμητα και μας ρώτησε τι κάνουμε και όταν είδε ότι και αυτός θα μπορούσε να συμμετέχει, πραγματικά τον κατέκλυσε ενθουσιασμός και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές συνταλλαγές και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Θεωρούμε λοιπόν και εμείς ότι πραγματικά οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν ποιες ευκαιρίες έχουν στη διάθεσή τους, τι μπορούν να κάνουν. Τι δυνατότητες τους δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνατότητες συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα. Μας ρωτήσατε επίσης πώς μπορούμε εμείς να προωθήσουμε περισσότερο την Ευρώπη. Μα νομίζω ότι η λέξη κλειδί εδώ πέρα είναι η κινητικότητα. Δεν μπορούμε να διδάξουμε, να μάθουμε στους νέους τι είναι η Ευρώπη αν οι νέοι δεν πάνε στην Ευρώπη, αν οι νέοι δεν ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Σαφώς μπορούμε να δώσουμε κάποια καθοδήγηση στα πλαίσια ενός, ε, στα πλαίσια της αίθουσα, στα πλαίσια του σχολείου βασικά. Πολύ συχνά όμως οι μαθητές δεν θα πρέπει να είναι απλώς παθητικοί δέκτες στα πλαίσια ενός μαθήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουν σαφώ κάποια πράγματα για την Ευρώπη στο σχολείο, αλλά θα πρέπει να βγουν και εκτό τάξη στη συνέχεια και να βιώσουν η δίσόμαση την Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας δώσετε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες προκειμένου και στο μέλλον να κάνουμε τέτοια project και ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει πολύ σύντομα. Θέλουμε να προωθήσουμε την εκπαίδευση, θέλουμε να προωθήσουμε την κατάρτιση και θέλουμε να τροποποιηθεί όμως και η μέθοδος εκπαίδευσης. Κύριε Γραμματικάκη, όταν σχεδιάσαμε το project αυτό, αντιμετωπίσαμε και οι ίδιοι κάποια προβλήματα. Καταφέραμε λοιπόν να αποφεληθούμε πάρα πολύ και εμεί οι ίδιοι από το ίδιο το project αυτό, ενώ το σχεδιάζαμε. Δηλαδή, ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε τι περιμένουν από εμά οι υπόλοιποι νέοι, γιατί και εμείς ακριβώς εκείνη την κατάσταση βρισκόμασταν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις αυτές, σας ευχαριστούμε επίσης και για τις αρχικές σας παρουσιάσεις. Μπορείτε να μείνετε τώρα μαζί μας αν θέλετε και για το υπόλοιπο της συνεδρίασης και μάλιστα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και για το πρόγραμμα Erasmus Plus από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι και το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη θα αναφερθούμε στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο Erasmus Plus που καλύπτει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση και τον αθλητισμό. Το Erasmus Plus αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της προηγούμενης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγκρίθηκε το νέο αυτό πρόγραμμα στα τέλη του 2013 και το Erasmus Plus θα διαρκέσει 7 χρόνια από το 2014 δηλαδή ως το 2020. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου χρόνου εκτέλεσης εφαρμογής αυτού του, του προγράμματος και θεωρώ την κατάλληλη στιγμή να κάνουμε έναν απολογισμό του πρώτου αυτού έτους. Πόσο μάλλον που ακούσαμε ότι έχουμε κάποια ανησυχητικά μηνύματα, καθότι υπάρχουν κάποιες περικοπές ή αδυναμίες καταβολής πληρωμών για το Erasmus+. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της μονάδας ECAC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα είναι σε θέση να μας ενημερώσει για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και ιδίω θα μας ενημερώσει για τις δημοσιονομικές περικοπές, δημοσιονομικές επιπτώσεις του προγράμματος αυτού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα σας κάνω μια σύντομη εισήγηση για το θέμα θα σας θυμίσω καταρχήν τι είναι το πρόγραμμα γιατί πολλοί είναι καινούργοι οι βουλευτές εδώ στην Επιτροπή και δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει το πρόγραμμα. Και μετά θα περάσω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και τι μάθαμε από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του. Το βασικό στοιχείο του Erasmus Plus είναι ότι προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε και παλαιότερα προγράμματα του Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus και άλλα μικρότερα και να τα συσσωματώσουμε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με βάση τρεις κύριες δραστηριότητες. Μία προφανής είναι φυσικά η κινητικότητα, αλλά Υπάρχουν και τα σχέδια συνεργασίας καθώς και η στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις. Κάτι που θέλαμε να πετύχουμε με το νέο πρόγραμμα ήταν περισσότερη αποτελεσματικότητα και γι' αυτό μειώσαμε ορισμένες δραστηριότητες και δράσεις και στοχεύσαμε σε πιο σημαντικές και μεγαλύτερες. Με ιδιαίτερη έμφαση στο τι κάνει κανείς και όχι στο ποιος είναι. Επίσης προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τη σύνδεση μεταξύ των στόχων που έχουμε στην, στον της παιδείας ας πούμε με τα προβλήματα των νέων και επίσης θέλαμε να διασφαλιστεί ότι θα υπήρχε καλύτερη πληροφόρηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Αυτές ήταν μερικές από τις αρχές. If we look at Το πρώτο κύριο στοιχείο η κινητικότητα. Βλέπετε εδώ λίγο, σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες τι δραστηριότητες στηρίζουμε. Για μεμονωμένους ε, υποστηρίζουμε την μετεκπαίδευση τους, την επαγγελματική τους μετεκπαίδευση για ήδη εργαζόμενους αυτά που βλέπετε εδώ. Μια αλλαγή με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι κάθε μεμονωμένη ατομική κινητικότητα πρέπει τώρα να συμπεριλαμβάνεται στην γενικότερη θεσμική προσέγγιση. Μέσω κάποιου οργάνου δηλαδή, όχι κανείς από μονομένα. Άλλη δραστηριότητα είναι τα κοινά προγράμματα μάστερ. Αυτό υπήρχε και υπό τον Έρασμος Μούντους είναι προγράμματα συνεργασίας πολλών εθνών και πανεπιστημίων όπου καθορίζονται κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, φοιτητικά δάνεια. στα οποία προσθέτουμε και μια εγγύηση, ένα σύστημα εγγύησεων για την μεγαλύτερη εκπαιδευτική κινητικότητα των φοιτητών σε επίπεδο μάστερ. Δεύτερη κύρια δραστηριότητα είναι η συνεργασία που θέλουμε να στηρίξουμε για την καινοτομία, δηλαδή για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πάλι. Έχουμε τις λεγόμενες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις σε συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων και κρατών και δύο πιο ειδικευμένες δράσεις τις λεγόμενες συμμαχίες γνώσης και συμμαχίες τομεακών προσόντων. που συνδέονται ιδιαίτερα με την ε, σχέση με τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε στον κάθε τομέα ας πούμε τι προσόντα λείπουν και προσπαθούμε να τα χορηγήσουμε από τα πανεπιστήμια. Αυτά είναι πιο μεγάλων διαστάσεων προγράμματα βέβαια. Στην πράξη, κάτι για το οποίο μιλούν πολλοί είναι οι προϋπολογισμοί, ο προϋπολογισμός μας. Με την υποστήριξή σας καταφέραμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό μας κατά 40% σε σχέση με τον προηγούμενη επταετή περίοδο. Το συνολικό ποσό για τα επταετή περίοδο λοιπόν είναι εδώ. Από το κεφάλαιο 1α, δηλαδή την αναπτυξιακή πλευρά του προϋπολογισμού και ένα μικρότερο τμήμα από εξωτερικά όργανα όπως το εργαλείο διεύρυνσης κλπ. Εδώ βλέπετε μία απλή γραφική παράσταση για τις δαπάνες της επταετούς περίοδους. Αυτή η 40% αύξηση της επταετούς περίοδου σε σύγκριση με την προηγούμενη επταετή περίοδο μας επιτρέπει να έχουμε έναν προϋπολογισμό που είναι σχεδόν διπλάσιος θα είναι διπλάσιο το 20 από ό,τι τώρα. Φτάνουμε τα 3 δισεκατομμύρια το 20 δηλαδή και τώρα είναι περίπου 1,5 λίγο παραπάνω. Δισεκατομμύρια μάλλον. Σημαντική αύξηση λοιπόν, αλλά επίσης βλέπετε ότι αρχίζουμε αρκετά χαμηλά. Αν προσθέταμε και το 13 θα βλέπατε ότι δεν είναι πολύ ψηλότερο από το 14, το 14 όχι πολύ ψηλότερο από το προηγούμενο κλπ. Η αύξηση αρχίζει από το 16 και μετά και ύστερα αυξάνεται γεωμετρικά τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια του προγράμματος. Μια ιδιαιτερότητα του νομικού υποβάθρου για το έρασμος πλούς είναι ότι υπάρχουν ορισμένα ποσοστά για την κατανομή του προϋπολογισμού του. Σε συζήτηση με εσά και με τα κράτη-μέλη καθορίστηκαν αυτά τα ποσοστά. Βλέπετε λοιπόν ανατομέα τα ποσοστά και ανακύριες δραστηριότητες. Είναι πολύπλοκο το σύστημα, ας πούμε, λέει ότι 77,5% του προϋπολογισμού πρέπει να αφιερώνεται στην μετεκπαίδευση και την παιδεία και μικρότερα ποσοστά σε άλλα στοιχεία του προγράμματος. Και τώρα μέσα σε αυτό το θέμα της παιδείας υπάρχουν και άλλες υποκατανομές. Ένα τρίτο του συνολικού, 33% τουλάχιστον δηλαδή, αφιερώνεται στην ανώτερη εκπαίδευση. Όχι μόνο μετεκπαίδευση και γενικότερη παιδεία. Αυτά είναι οι παράμετροι που πρέπει να γνωρίζουμε όταν θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Επίσης για τις δραστηριότητες κάτω, στο κάτω μέρος βλέπετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι για την κινητικότητα. 3,5% και στη συνεργασία και μετά η στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις σε σταθερό ποσοστό 4%. Κάτω-κάτω βλέπετε κάποια ελαστικότητα στους αριθμούς ανατομέα, 5% ελαστικότητα. Προηγουμένως είχαμε δει ότι το συνολικό ποσό των, το συνολικό ποσό των 7 ετών, γιατί για το σύνολο μιλάμε, όχι για κάθε χρόνο, αν βλέπετε λοιπόν εδώ 10% για την νεολαία, έχουμε 14,5 δισεκατομμύρια σύνολο για τα 7 χρόνια, 1,4 δηλαδή για την νεολαία, συν πλην 5%. Αυτό είναι η ελαστικότητα που σας έλεγα. Άλλο σημαντικό που πρέπει να ξέρετε αν συζητάτε τον προϋπολογισμό είναι ότι ο προϋπολογισμός του Erasmus Plus έχει τέσσερις θέσεις στον προπολογισμό του. Μία θέση τη μεγαλύτερη για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, μία για την νεολαία, μία για το Ζαν Μονέ και μία για τον αθλητισμό. Τα δύο τελευταία είναι μικρότερα βέβαια. Να θυμάστε λοιπόν ότι αν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα αυτές οι τέσσερις θέσεις του προϋπολογισμού είναι σημαντικές. Υπάρχει και μια άλλη θέση τεσσερα στον τμήμα τέσσερα μάλλον, για ειδικά λειτουργικά προγράμματα γειτονία, γειτονία κλπ. Για τη διαχείριση σας είπα ότι γίνεται από τις εθνικές υπηρεσίες και από την ΕΑΚΕΑ, κυρίως από τις εθνικές 80% και 20 περίπου από την ΕΑΚΕΑ. Ε, πολύ μικρό ποσοστό κατευθείαν από την Κομισιόν. Άλλο σημαντικό στοιχείο που άλλαξε ήταν μια απλοποίηση που προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσω μεγαλύτερης κατανομής ε, του κόστους αναμονάδα. Πράγμα το οποίο μειώνει και τον κίνδυνο λαθών ε, τι μάθαμε από το φετινό έτος. Το 2014 ήταν ο πρώτος χρόνος του προγράμματος και γι' αυτό κάθε αρχή και δύσκολη. Είπαμε ότι το κυριότερες δραστηριότητες γίνονται από εθνικές υπηρεσίες, 60 τέτοιες υπάρχουν. Τις εξετάσαμε όλες για να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργούν σωστά οι έλεγχοι αυτοί βέβαια ήταν ελαφρότεροι αν είχαν ξαναγίνει και στο παρελθόν από ότι αν για πρώτη φορά. Έχουμε γράψει νέους κανόνες, το λεγόμενο Program Guide, νέο λογισμικό για το πρόγραμμα και εντωμεταξύ συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε και τα παλαιότερα προγράμματα, τα τελευταία χρόνια των προηγουμένων περιόδων δηλαδή. Βέβαια υπήρξαν και μερικά προβλήματα φυσικά για την αρχή. Η εφαρμογή ήταν χαμηλότερη, αργότερη φέτος από ότι τον πρώτο έτος του προηγούμενου προγράμματος Άρα μερικές προθεσμίες δεν έγιναν ακριβώς σεβαστές, αλλά ήδη στο δεύτερο χρόνο θα υπάρξει ο κανονικός ρυθμός εφαρμογής όπως για το προηγούμενο πρόγραμμα. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα είναι αυτό που λέμε πληθωρισμό των, του μεγέθους των προγραμμάτων, δηλαδή έχουν την τάση να μεγαλώνουν άρα μπορούμε να επιλέξουμε λιγότερα. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είναι απαραίτητες οι διαστάσεις ορισμένων προγραμμάτων και ότι δεν γίνεται απλώς υπερβολή, δεν γίνεται απλώς υπερβολή. Μερικά προγράμματα δεν άρχισαν ακόμα γιατί το νομικό υπόβαθρο εγκρίθηκε φέτος πολύ αργά δηλαδή για να εφαρμοστεί. Αλλά δεν θα χαθούν τα χρήματα, θα χρησιμοποιηθούν σε 6 χρόνια αντί για 7. Τα φοιτητικά δάνεια δεν άρχισαν ακόμα, ακόμα γίνεται η προετοιμασία. Και οι πρώτες δεσμεύσεις ή προβλέψεις υπάρχουν, αλλά οι πληρωμές αρχίζουν του χρόνου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε όλο τον προϋπολογισμό ή όλο το πρόγραμμα. Όλο τον προϋπολογισμό θα χρησιμοποιήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί όπως σας έδειξα και πριν, ο προϋπολογισμός δεν είναι και τόσο ψηλός φέτος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες της χώρες μέλη γιατί είπαμε θριαμβευτικά ότι έχουμε 40% μεγαλύτερο προϋπολογισμό αλλά όχι από φέτος. Έπεσε λίγο ο ενθουσιασμός λοιπόν γιατί δεν δώσαμε πολύ περισσότερες πληρωμές ή πολύ περισσότερα προγράμματα. Σχετικά χαμηλές, χαμηλή ρυθμή επιλογών λοιπόν, αυτή είναι προκατρακτική αριθμή βέβαια. Βλέπετε χαμηλό αριθμό για την νεολαία αλλά αυτό θα αυξηθεί ακόμα. και η κύρια δράση 2 για τα σχολεία δεν είναι 10% ήδη αλλά 17%. Η ρυθμή αυτή επιλογής λοιπόν των σχεδίων δεν είναι πολύ ψηλή και αυτό πρέπει να το ξαναδούμε για το Erasmus Plus γιατί πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα για να ενδιαφερθούν αρκετοί. Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός του χρόνου θα μας βοηθήσει βέβαια και για αυτά. Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η έλλειψη πληρωμών Νομίζω δεν σας εκπλήσει, υπάρχει γενικά αυτό το πρόβλημα στην Ένωση. Στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν προβλέπονται επαρκείς πληρωμές από την αρχή. Αυτό φαίνεται από έναν αριθμό. Το 14 σε σύγκριση με το 13 οι δεσμεύσεις τα προγράμματα που μπορούμε να υπογράψουμε δηλαδή, είναι 9% παραπάνω από ότι το 13% ενώ για τις πληρωμές 13% λιγότερο από πέρυσι. Είναι λοιπόν σαφές ότι δεν έχουμε αρκετά κονδύλια για τις πληρωμές. Τι κάναμε λοιπόν για να το αντιμετωπίσουμε. Καθυστερήσαμε τις πληρωμές λιγάκι στην αρχή κάνουμε μία προκαταβολή, αυτές τις μειώσαμε για να μπορέσουμε να τους πληρώσουμε όλους λίγο λιγότερο βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελικά θα πληρώσουμε λιγότερα. Θα πληρώσουμε περισσότερα, αλλά ίσως πιο αργά. Και παρόλα αυτά, μας λείπουν λεφτά. Ξέρετε ότι ζητήσαμε 202 εκατομμύρια παραπάνω πληρωμές για φέτος σε έναν από τους αναθεωρητικούς προϋπολογισμούς. Και ήδη σήμερα 1η Δεκεμβρίου κάνουμε τις τελευταίες πληρωμές που έχουμε. Μετά από λίγες μέρες δεν θα έχουμε καθόλου λεφτά για πληρωμές. Αν δεν πάρουμε τα 202 εκατομμύρια λοιπόν που ελπίζαμε να είχαμε πάρει περίπου τώρα, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε για το υπόλοιπο μήνα. Τώρα, πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν οι φοιτητές και τα λοιπά. Αφού δουλεύουμε με το σύστημα των εθνικών υπηρεσιών, αυτές έχουν ακόμη λίγα αποθέματα για τον τελευταίο μήνα. Σημαίνει όμως ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να πληρωθούν πολύ νωρίς του χρόνου αν δεν πάρουμε τα 202 εκατομμύρια να τα πληρώσουμε από τον προπολογισμό μας το 15. Θα αρχίσουμε λοιπόν δημιουργώντας έλλειμμα στον προπολογισμό μας ή αυξάνοντας το χάσμα και το έλλειμμα, αυξάνοντας. Αφού δεν είχαμε και φέτος αρκετά χρήματα, δεν θα έχουμε αρκετά και του χρόνου. θα μεγαλώσει το χάσμα και τελικά τον επόμενο Δεκέμβριο θα είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι σήμερα. Δεν μπορώ να σας τα πω ακριβώς, αλλά ίσως το φθινόπωρο ήδη να υπάρξει το πρόβλημα. Σημαντικό λοιπόν θέμα για τη βιωσιμότητα του προγράμματος. Αν οι προϋπολογισμοί αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, θα αυξηθούν, αλλά δεν μπορούμε συνεχώς να προκαταβάλουμε και για τα επόμενα χρόνια, γιατί συνεχώς δεν θα υπάρχουν αρκετές πληρωμές σε σύγκριση με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Σημαντικό λοιπόν το θέμα. Ξέρω ότι θα μας υποστηρίξετε σε αυτό. Αλλά πρέπει και το Συμβούλιο να συμφωνήσει. Αυτά. Και φυσικά είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γλέζος πρώτος. Με ιδιαίτερη προσοχή επί 25 λεπτά περίπου παρακολούθησα την ανάπτυξη ενός φιλόδοξου σχεδίου, του φιλόδοξου σχεδίου Έρασμος και που έχει αρκετή επιχορήγηση άλλο αν παρουσιάζονται τα ειδικά προβλήματα ε, ίσπραξης των χρημάτων. Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι ένα. Με ποιο δικαίωμα αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον της νεολαίας χωρίς να συμμετέχουν οι νέοι που τους αφορά αυτούς τους ίδιους σε αυτή τη συζήτηση. Είχα την ευκαιρία προχθές Παρασκευή να προσκληθώ στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Λουξεμβούργου. Ένιωσα την μεγάλη και ιδιαίτερη συγκίνηση που νιώθω όπως στην πατρίδα μου την Ελλάδα έχω προσκληθεί και έχω μιλήσει σε πάνω από 400 σχολεία από τον Υπηαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο. Δεν έκανα εισήγηση, προσέξτε αυτό ειδικά το θέμα, δεν έκανα εισήγηση. Ζήτησα από τους μαθητές να ανταλλάξουμε απόψεις, να με ρωτήσουν και να ρωτήσω, να ρωτήσω και να με ρωτήσουν να αναπτυχθεί ένας διάλογος. Και το Προεδρείο που διεξήχθη, έκανε τη διεξαγωγή της συζήτησης αυτής ήταν μια κατάκτηση επίσης της δημοκρατίας. Το αποτελούσε η διευθύντρια του σχολείου, ο προσκεκλημένος που ήταν η αφεντιά μου και ένας μαθητής εκλεγμένος από τους ίδιους τους μαθητές. Όταν μάλιστα ξεκινήσαμε, διήθυνε αυτός πρώτος στη συζήτηση και είπε να κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση. Του είπα ακόμα δεν πήρε την εξουσία και θες να την εκμεταλλευτείς και κάτω από την επιδοκιμασία όλων αφέθηκε να κάνει το ερώτημα τελευταίος. Ήταν ένα μάθημα δημοκρατίας. Υπήρξε ένας γόνιμος διάλογος, αρκετά σημαντικός και αναρωτιέμαι το πρόγραμμα Έρασμους, όπως και η προηγούμενη συζήτηση, την οποία παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή, είναι ένα πρόγραμμα τι, για τους νέους ή επιβολής των απόψεών μας στους νέους. Αυτό είναι το ερώτημα. Το μόνο δικαίωμα που έχουμε δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση να μεταφέρουμε τις γνώμες μας τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας στους νέους, αλλά όχι ανεξέλεκτα. Οι ίδιοι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν στον τρόπο της απόκτησης αυτής της εμπειρίας. Δεν ξέρω, Κι άλλες φορές έχω μιλήσει εδώ, νομίζω ότι μιλάω ως φωνή εν Ελπίζω αυτή τη φορά κάποιοι να μ' ακούσουν, έστω και οι Κύπριες που βρίσκονται μπροστά μου, οι οποίες δυστυχώς δεν μίλησαν την ελληνική γλώσσα, αλλά μίλησαν την αγγλική. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Τους επιβάλαμε να μιλήσουν την αγγλική. Όχι με επιβολή έτσι, είναι και άλλος τρόπος επιβολής. Δηλαδή, πιο καλύτερα θα είναι για σας να μιλήσετε στα αγγλικά για να δείξετε ότι κατάχετε και την αγγλική γλώσσα. Καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο, δηλαδή με, με ποιο ε, δέλεαρ τις πείσαμε να μην μιλήσουν στη γλώσσα τους. Πρωτοφανέρο το γεγονός. Και ευτυχώς που είναι μπροστά μου και μ' ακούνε και ελπίζω να μην το επαναλάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Κυρία έχει το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιό και πρέπει να παραδεχθώ ότι με εκπλήσουν όχι μόνο οι αριθμοί που άκουσα, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιες συζητήσεις που έπρεπε να είχαμε εδώ δεν έγιναν. Στην απόφαση, αν δεν κάνω λάθος που είχαμε λάβει, είχαμε πει ότι στην Επιτροπή μας είχαμε αποφασίσει να διατηρηθούν κάποια παλιά προγράμματα με τον τίτλο που είχαμε. Δεν τα αναφέρεται Έρασμος, Youth in Action, Leonardo, Da Vinci. Ήτανε προγράμματα βασικά και είπαμε ότι θα πρέπει να μην τους αλλάξουμε όνομα. Δεν τα άκουσα να τα αναφέρετε. Τώρα μιλάτε μόνο για τρεις δράσεις, τρία προγράμματα. Εκπλήσωμε, λοιπόν. Και είμαι και δυσαρεστημένη. Διότι ήταν πολύ σημαντικό το θέμα και με δυσαρεστεί επίσης το ότι πρέπει να διαπιστώσουμε ακόμη μια φορά ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των πιστώσεων υποχρεώσεων και των πληρωμών. Και όπως είπατε, οι εθνικοί οργανισμοί έχουν περιθώριο. Ακούστε, εγώ όσον αφορά τη δικό μας τον οργανισμό, τον ε, ε, γερμανικό, ξέρω ότι δεν θα έχουμε SAE περιθώριο λιγμών, δεν θα έχουμε πλέον χρήματα. Και του χρόνου πάλι στην ίδια κατάσταση θα είμαστε. Από την αρχή του χρόνου. Δεν θα διαπιστώσουμε το Δεκέμβριο ότι δεν έχουμε χρήματα. Ήδη από το Σεπτέμβριο θα το δούμε. Και έτσι κανένας εθνικός οργανισμός δεν θα είναι σε θέση να συνεισφέρει θετικά. Συν 9% είπατε. Αυτό σημαίνει μείον 13% στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιου είδους θέματα. Και βεβαίως ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση. Μας λένε από τη Γερμανία ότι κυρίως στα θέματα ε, συνεργασίας μεταξύ σχολείων στα πλαίσια του προγράμματος Κομένιους και εξαιτία τεχνικών αλλαγών που έγιναν υπευλήθησαν πολύ λιγότερες αιτήσει από ό,τι στο παρελθόν. Πράγμα που δεν οφείλεται μόνο σε αλλαγέ τεχνικού περιεχομένου ή σε θέματα αλλαγή του εντύπου για την ε, υποβολή Υπάρχει μεγάλο ποσοστό απόρριψη των σχεδίων που υπεβάλλονται. Θα ήθελα εγώ αυτές οι εταιρικέ σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ σχολείων να ενθαρρυνθούν και να χρηματοδοτηθούν περισσότερο από του χρόνου, δεδομένου ότι αποτελούν ένα από τα στοιχεία κλειδιά του προγραμματό μα και δεν μπορούμε να δεχθούμε να υποβληθούν πολύ λιγότερες αιτήσει από ότι πέρσι ο στόχος μας ήταν να απλοποιήσουμε τα πράγματα ώστε οι διατυπώσεις για την υποβολή αιτήσεων να είναι πιο απλή, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα διάφορα έντυπα είναι πολύ πιο δύσκολα να τα συμπληρώσει κάθε σχολεία, στα πλαίσια του κομμένιους και πάλι επαναλαμβάνω. Άρα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε για να αλλάξουν τα πράγματα και του χρόνου να υπάρχουν περισσότερα ε, σχέδια κομμένιους που θα θα κάνουμε την έρευνά μας και για τα υπόλοιπα, αλλά αυτά είναι αυτά που θέλω να πω ως πρώτες παρατηρήσεις για το κομμένιου σε σχέση με το σύνολο των κονδυλίων που διατίθενται και με τις αιτήσει που υποβάλλονται. Κυρία Βαρέ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Κάμερβέρτη. Πραγματικά και εμένα μου έκανε εντύπωση ο πίνακας αυτός που μας δείξατε, καθώς επίσης και τα ποσοστά για ορισμένα σχέδια. Πραγματικά ενοχλούμε πάρα πολύ όταν βλέπω ότι ε, έχουμε κάποια αριθμητικά δεδομένα ιδιαίτερα χαμηλά όσον αφορά την χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων. Και λυπάμαι που δεν βλέπω κάποια προγράμματα ιδιαίτερα γνωστά, να έχουν διατηρήσει δηλαδή την αρχική του ονομασία. Πραγματικά αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Σε άλλες περιπτώσεις μας είπατε ότι για κάποια σχέδια είχατε κινητοποίηση 100% από την άλλη όμως μας είπατε ότι απορρίψατε και κάποια σχέδια, κάποια προγράμματα. Για ποιο λόγο έγινε αυτό μπορείτε να μας το πείτε. Για τυπικούς λόγους δεν σας δόθηκε απαραίτητη ενημέρωση, δεν υπήρχε απαραίτητη χρηματοδότηση. Για ποιο λόγο ένα τέτοιο υψηλό ποσοστό απόρριψης. Όσον αφορά τώρα την υλοποίηση, την εφαρμογή από τις εθνικές υπηρεσίες. Ακούω πολλά και διαφορετικά πράγματα από τι εθνικέ υπηρεσίε για το αν υφίστανται ή όχι προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω από εσά τι πραγματικά συμβαίνει. Μπορείτε, αν μη τι άλλο, να μα υποβάλλετε μια έκθεση υλοποίηση εφαρμογή για το Erasmus Plus, μια επίσημη έκθεση. Μας δείξετε επίσης μια γραφική παράσταση με μια καμπύλη, και μας είπατε ότι μεσοπρόθεσμα έχει εντοπίσει ήδη κάποιες περιόδους όπου μπορεί να έχουμε προβλήματα χρηματοδότησης. Μας είπατε επίσης ότι ε, αρχικά θα έχουμε κάποια προβλήματα, μια κάποια στασιμότητα στη χρηματοδότηση, αλλά έπειτα αυτό θα αντισταθμιστεί από απότομη αύξηση της χρηματοδότησης. Ποιο είναι ακριβώς το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνουμε όμως αυτή τη στιγμή. Η αύξηση αυτή τη χρηματοδότηση μπορεί να επέλθει μετά από δύο-τρία χρόνια. Αν όμω έχουμε καταναλώσει ήδη όλο τον προπολογισμό μα μέχρι τότε, τι θα κάνουμε, πώ θα καλύψουμε δηλαδή το ενδιάμεσο διάστημα. Μήπω βρεθούμε κάπω εκτεθειμένοι. Και α μην ξεχνάμε ότι τα πράγματα μπορεί να αποβούν ακόμα χειρότερα στο μέλλον. Τα κράτη-μέλη ενδεχομένω να κάνουν ακόμα περαιτέρω περικοπέ στο μέλλον. Τι θα κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε έναν κάποιο σχεδιασμό, μια κάποια βεβαιότητα, μια κάποια ασφάλεια για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του ή μήπως θα καταφέρουμε τελικά να χρηματοδοτήσουμε μόνο την αρχική του φάση χωρίς να καταφέρουμε να καλύψουμε το σύνολό του. Καταλαβαίνετε ότι ε, δεν δίνουμε επίση τις απαραίτητες διασφαλίσεις και στους φοιτητές εκείνους που θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα αυτά για να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Το είχαμε τονίσει αυτό και στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος του Εράσμους και βλέπουμε πάλι ότι τέτοια προβλήματα προκύπτουν τώρα. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες λοιπόν και δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στις πληροφορίες αυτές. Έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια νέα διάρθρωση επίσης. Μέρος του προγράμματος Εράσμους εμπίπτει και στην αρμοδιότητα της κυρία Τάισεν, τυπικά τουλάχιστον. Ξέρετε, το πρόγραμμα Λεωνάρντο Νταβίντσι έχει να κάνει με την επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα τη κυρία Τάισεν. Όσον αφορά τα ζητήματα εκπαίδευση, παιδεία, αυτό εμπίπτει προφανώ στον τομέα του πολιτισμού και τη παιδεία, αλλά αρμόδιο ήταν ο Επίτροπο Ναύρατσιτ. Συγκεκριμένα πώ θα υλοποιηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά τα προγράμματα, ποιο θα είναι υπεύθυνο για ποιο πρόγραμμα υφίσταται ή όχι κάποιο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών αυτών επιτρόπων. Θα ήθελα επίση να γνωρίσω η καθημερινή βάση πώ οργανώνεστε, όχι μόνο σε μακροχρόνιο επίπεδο. Κυρία Τρούγκελ, θα ήθελα πραγματικά να επικρίνω το Συμβούλιο όσον αφορά το ζήτημα των πληρωμών. Έχουμε πλέον απτά αριθμητικά δεδομένα. Αν έχουμε μία μείωση 13% φέτο, αυτό αντιτίθεται στα όσα πολιτικά μα υποσχέθηκε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό το Κοινοβούλιο. Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ αρνητικό δίνει μια πολύ αρνητική εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικρίνουμε, να αποδοκιμάσουμε το Συμβούλιο πολύ χειρά, πολύ έντονα, γιατί ουσιαστικά με τη δράση του βάλει κατά της αξιοπιστία... των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεύτερον, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, τι θα γίνει με τις παλαιότερες ονομασίες των προγραμμάτων. Σαφέστατο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε πει ότι θέλουμε να διατηρηθούν τα ονόματα αυτά, καθότι είναι πολύ πιο γνωστά από τα νέα αυτά ονόματα στους ε, ετούντες. Τώρα, όσον αφορά τον οδηγό για τους ετούντε, για ποιο λόγο δεν έχει μεταφραστεί αυτός ο οδηγός σε όλες τις γλώσσες. Και όσον αφορά την ιστοσελίδα σας, για ποιο λόγο είναι μόνο στα αγγλικά η νέα σας ιστοσελίδα και αυτό δεν είναι πολύ φιλικό για το χρήστη όπως το καταλαβαίνετε και κάποιες καταγγελίες, κάποια παράπονα που έχουν φτάσει σε μένα. Υπάρχουν σχολεία, πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία επιθυμούν να κάνουν αίτηση για τα προγράμματα αυτά, αλλά έχουν κουραστεί πάρα πολύ από το σύστημά σας. Λένε ότι το όλο σύστημα επιβολής αίτησης γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, λένε τους ζητάτε όλο και περισσότερο αριθμητικά δεδομένα και ουσιαστικά συμβάλλεται στο να αποθαρρύνετε πάρα πολλούς ε, υποψηφίους. Θα ήθελα εγώ αντίθετα να είχαμε πολύ πιο εύκολο και απλό σύστημα για τις αιτήσει, προκειμένου να κινητοποιηθούν όλο και περισσότεροι νέοι, όλο και περισσότεροι δικαιούχοι να κάνουν αίτηση για τα προγράμματα αυτά. Σας παρακαλώ πολύ Ας το λάβετε αυτό υπόψη σας. Πολλές φορές πολύ φοβάμαι ότι με το νέο αυτό σύστημα, το πολύπλοκο σύστημα αιτήσεων, τελικά αποθαρρύνεται τους υποψηφίους. Ο κύριος Μοργκάνο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίασή του και όπως είπαν και οι προλύσαντες θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο ερωτήματα. Βλέπουμε ότι οι προβλέψεις όσον αφορά τις πληρωμέ αντιστοιχούν σε αυτή την καμπύλη όπου θα διπλαστεί τελικά ο προπολογισμό, όπως είπατε, το 2020. Τι θα γίνει όμως με τον προπολογισμό που θα έχουμε το 2016, ποιες εγγύσεις έχουμε αυτή τη στιγμή βράχει πρόθεσμα έτσι ώστε το 2016 να μην έχουμε μείωση στις πληρωμές. Δεύτερη ερώτηση. Σε σχέση με τους πόρους αυτούς οι οποίοι δεν αρκούν, όπως είπατε, θα ήθελα να γνωρίζω πόσο κοστίζει το όλο σύστημα το οποίο εσείς έχετε θεσπίσει. Πόσο δαπανηρό ενδεχομένως να είναι το σύστημα αυτό και πόσο επιβαρύνει τη χρηματοδότηση των τεσσάρων προγραμμάτων στα οποία αναφερθήκατε. Και κάτι ακόμα. Όταν θα έχετε όλα αυτά τα διαθέσιμα αριθμητικά δεδομένα, γιατί μας είπατε ότι αυτή τη στιγμή μας παρουσιάζεται μόνο μερικά μόνο προκαταρακτικά στοιχεία. Θα θέλαμε κι εμείς τότε να μας δώσετε μια οριστική τελική έκθεση που θα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα δεδομένα και θα μας επιτρέπει και σε εμάς να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Mrs. and then one more question, Helga Trupa. But, uh... κυρία Τρούπερ, μια ερώτηση, αλλά σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι, γιατί έχουμε συνάντηση των συντονισμών. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι που έχουμε αυτή την συζήτηση εδώ. Πρέπει να πούμε ότι το ο έρασμος ως πρόγραμμα είναι ένα οικονομικό μέσο για να υλοποιήσουμε κάποιους στόχους. Και αν δεν υλοποιηθεί σωστά το πρόγραμμα αυτό, δεν θα υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Είναι εύκολο να το εξηγήσει κανείς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Εάν θέλουμε όντως να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2020, θα πρέπει το Erasmus Plus να το χρησιμοποιήσουμε ως το μέσον που θα μας επιτρέψει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι διαπίστωσα ότι υπάρχουν προβλήματα στους κανονισμούς για την σύναψη εταιρικών σχέσεων, διότι οι διάφοροι οργανισμοί δεν μπορούν να περιορίσουν τα κονδύλια που χορηγούνται για κάθε σχέδιο. Στην προηγούμενη περίοδο μπορούσε κανείς να θέσει ανώτατο όριο στα προγράμματα, αλλά τώρα άλλαξε ο κανονισμός και υπάρχουν προβλήματα. Δεδομένου ότι πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια διαφορετικά. Ευχαριστώ, κυρία Τρούπελ. Μία συμπληρωματική ερώτηση. Τι οικονομική εγγύηση δίδεται για τους φοιτητές. Ο κύριος Μαραγάλια τελευταίος. Γεια σας. Πιστεύω ειλικρινά ότι είχε την ατυχία εκπρόσωπος της Επιτροπής σήμερα να μιλήσει μετά από τους νέους που κέρδισαν το βραβείο του Κάρλο Μαρλού. Διότι αν δούμε τι λένε οι νέοι, ποιες είναι οι δεσμεύσεις τους και τι μπόρεσαν να κάνουν ε, με πολύ λίγα χρήματα, έτσι όπως βλέπουμε να γίνονται τα πράγματα με την Κομισιό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι νέοι φεύγουν από εδώ με την εντύπωση ότι τους απονέμουμε ένα βραβείο, αλλά τους τιμωρούμε συγχρόνως. Δεν υπάρχει λοιπόν συνεκτικότητα σε αυτό που κάνει η Κομισιόν και θα πρέπει να σκεφτεί το εξή. Πώ αυτή την συγκεκριμένη στιγμή θα μπορέσει στα πλαίσια μιας νέας οικονομικής πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, ποιο ρόλο θέλει να έχει η παιδεία, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση. Δηλαδή, αυτό που είναι βασικό είναι να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν σωστά τα προγράμματα αυτά, κυρίως στα πλαίσια του σε επαγγελματική κατάρτισης και πώς θα πρέπει να δώσουμε μία νέα πνοή σε αυτά τα προγράμματα. Ακούγοντας τι έχουν να πούνε τα νέα παιδιά για την κινητικότητα και πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την κινητικότητα μεταξύ άλλων, να το κάνουμε. Και βεβαίως το εράσμος, ποια σημασία έχει. Να μπορέσει να προσεγγίσει και να κάνει να υποφεληθούν όλο και περισσότερα νέα παιδιά που σπουδάζουν. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νότς να απαντήσει την ερώτηση τώρα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω κάποιες ερωτήσεις. Όσον αφορά τους τίτλους των προγράμματος, υπάρχουν. Δεν τα χρησιμοποίησα ακόμη, το ονομασία του προγράμματος. Γιατί. Γιατί καμιά φορά είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιεί κάποια ονομασία ε, πιο γενική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα γνωρίζετε τα προγράμματα. Ξέρετε τι σημαίνει και σε ποιον εφαρμόζεται το Λεωνάρντο, σε ποιον το τα κτλ. Χρησιμοποίησα λοιπόν ε, για τον κάθε κλάδο γενικότερες παρατηρήσεις χωρίς να πω ποιο είναι ο τίτλος κάθε προγράμματος όπως σωστά επισημάνατε. Υπήρχαν κάποια σχόλια που αφορούν επίσης τον προπολογισμό, τα κονδύλια. και το περίγραμμα, το προφάιλ αυτό. Δεν είναι κάτι το που αφασίζει μόνο η Κομισιό, είναι κάτι που είχε αποφασιστεί στα πλαίσια του πολιετού χρηματοδοτικού προγράμματος, στα πλαίσια των αποφάσεων που έχει λάβει και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όντως, για το 2016 προβλέπεται μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν αλλαγές στα πλαίσια της αναθεώρησης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται σωστά και αποδίδουν, έχουν αποτελέσματα προγράμματα κατά τη διάρκεια της ε, ε μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης. Το ίδιο συνέβη και στο μέσο της προηγούμενης πολιετούς περίοδου και αν αποδειχθεί ότι ανταποκρίνεται στην Ευρώπη στις ε, δυνατότητες ανάπτυξης στην αθεώρηση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα δούμε πώς θα συνεχιστούν. Αυτό θα γίνει στο 2016, επαναλαμβάνω, αλλά θα πρέπει να επαγρυπνούμε, είναι σαφές. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί αυξηθεί ε, πολύ το συνολικό ποσό το οποίο δίνεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Ναι, αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, ανάλογα. Και με τις οργανώσεις και τους υποψηφίες. Ε, έχουμε προσπαθήσει να απλοποιήσουμε τα πράγματα αλλά ξέρουμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και κίνητρα, να υπάρχει ενδιαφέρον για αυτά τα προγράμματα. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες αιτήσει οι οποίες είναι αντιμαχόμενες, αντιφατικές. Για να δώσουν περισσότερα χρήματα πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε εκθέσεις αναφοράς για να ξέρουμε τι σημαίνει στην πράξη. Ζητούμε από όλους όσοι συμμετέχουν σε τέτοιου προγράμματα και περισσότερο από το παρελθόν όσοι συμμετέχουν να μας κάνουν αναφορές για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, όταν δεν είναι χρήσιμο δεν ζητούμε να γίνονται τέτοιου είδους αναφορές. για τις δαπάνες ε, ταξιδίου. Έχουμε θεσπίσει το σύστημα της ε, μονάδας ε, αντικαταβολής για τα ταξίδια, οπότε είναι πιο απλό το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητούμε, για να ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα κάθε προγράμματος, περισσότερες εκθέσεις αναφοράς. Γι' αυτό το reporting, η αναφορά δηλαδή, θα πρέπει να, είναι, να γίνεται με απλό τρόπο και να αποφεύγουμε ε, να ζητούμε και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Ήδη στις αιτήσει παίρνουμε κάποιες ε, πληροφορίες που μας επιτρέπουν να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ένα πρόβλημα. Αλλά όντως το reporting αυτής της αναφορές είναι ένα άχθος για τους στοιχείους, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης γίνανε κάποιες παρατηρήσεις. για την ε, έλλειψη αρκετών προγραμμάτων ε, ε, συνεργασίας των σχολείων στα πλαίσια του Κομίνιους. Θα πρέπει να το εξετάσουμε εκ του σύνεγγης το θέμα αυτό, γιατί πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος οι εθνικοί οργανισμοί δεν χρησιμοποίησαν αρκετά την δυνατότητα που έχουν να υποβάλουν ανάλογα με τα κονδύλια που είχαν στην διάθεσή τους τα κατάλληλα προγράμματα. Και θα πρέπει να υπάρχει λογική μεταξύ των κονδυλίων που διαθέτει ο καθένας και αυτών που ζητάνε κάτι στα πλαίσια του προγράμματος, να μην ξεπερνιούνται κατά πολύ τα κονδύλια. Διότι αν ξεπερνιόνται τα επιτρεπόμενα κονδύλια σε κάθε προϋπολογισμό, το, επιλέγονται λιγότερα προγράμματα. Αυτό το συζητούμε με τους εθνικές οργανισμούς και προσπαθούμε να τους κάνουμε να συμμετέχουν περισσότερο ώστε να μην παρουσιάζονται πολύ δαπανηρά προγράμματα ώστε να περνούν λίγα και οι περισσότεροι να μένουν απ' έξω. Uh, Τώρα, η κυρία Κάμερβερτ ανέφερε το θέμα των προβλημάτων πληρωμής. Ξέρουμε ότι προς το παρόν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να καλύψουμε τις ανάγκες που μπορούμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Του χρόνου θα δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά, όπως είπατε, μπορεί να μην έχουμε χρήματα, να εξαντλήσουμε τους πόρους των διαθεσή μας και μετά το καλοκαίρι να χρησιμοποιήσουμε κάποια βοηθητικά κονδύλια, αλλά δεν είναι και αυτά ανεξάντλητα. Τώρα, κάποια ποσοστά που είπατε και το πώς επωφελούνται περισσότερο τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα ποσοτά του είναι πολύ περισσότερα δηλαδή στα πλαίσια των διαφόρων δράσεων. Γι' αυτό είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό τους, γιατί κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια τις τα ίδια πανεπιστήμια που υποβάλλουν αιτήσει. Και βεβαίως η κινητικότητα είναι κάτι που γίνεται μέσω θεσμών, μέσω πανεπιστημίων, ε, ιδρυμάτων. Δεν γίνεται ατομικά για τον καθένα. Στα σχολεία τα πράγματα είναι ε, διαφορετικά. Επίσης είπατε ότι στο παρελθόν οι φοιτητές, αν δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα, έπαιρναν ε, μικρότερο ποσό υποτροφίας. Τώρα τα αλλάξαμε τα πράγματα, διότι αναγγέλουμε εκ των προτέρων ποια είναι τα ποσά των υποτροφιών που δίδονται και δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Όπω είπατε βεβαίω τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λέτε. Δηλαδή αν μειωθεί το ποσό της υποτροφίας ίσως δεν θα μπορούν να σταλούν και τόσοι πολλοί φοιτητέ. Για να καλυφθούν δηλαδή όλες οι οικονομικές ανάγκες, άρα θα αποστέλλονται για το ίδιο ανώτερο ποσό, λιγότεροι φοιτητέ. Τώρα, η μείωση των πιστώσεων πληρωμών στα πλαίσια σε ποσοστό 13%. Στα πλαίσια του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί στο παρελθόν, δεν έγινε φέτος. Οι μεταφράσεις φτάνουν. Συνεργαζόμαστε με όλους τους εθνικούς οργανισμούς ώστε όλα τα φυλάδια, τα έντυπα, τα σχετικά να μεταφράζονται στη μητρική γλώσσα του καθενός. Αλλά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα, το σύστημα εγγύησης για τα δάνεια που δίδονται, που χορηγούνται στους φοιτητές, ελπίζουμε ότι οι συμφωνίες θα υπογραφούν φέτος με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και θα αρχίσει η χορήγηση αυτού του είδους των δανείων για τους φοιτητές από του χρόνο. δαπάνες προσωπικού. Διοικητικές. Υπάρχει ένα νοτοτόριο που προβλέπεται στη νομική βάση. Το νοτοτόριο για διοικητικές δαπάνες είναι 1,9% για, διοικητικές, ε, για δαπάνες ε, διοικητικών περίπου 3%. Καταλαβαίνετε ότι στην αρχή όταν θεσπίζεται ένα νέο σύστημα υπάρχουν πολλές δαπάνες και για τα συστήματα πληροφόρησης και κάθε χρόνο θα μειώνονται αυτές οι δαπάνες. Δεν είναι δαπάνες που ανολογικά θα αυξάνουν κάθε χρόνο. Συνεχίζει η εφαρμογή. Δεν μπορώ να σας δώσω τα τελικά στοιχεία θα συνεχιστεί και στις αρχές του επομένου έτους για διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν χρονική διάρκεια 2-3 ετών, άρα τα τελικά δεδομένα θα τα έχουμε στο πέρος, πέρας κάθε προγράμματος. Περίπου του χρόνου το φθινόπερο, περίπου θα, θα έχουμε μία σφαιρική εικόνα για τα προγράμματα και τις δαπάνες. Επίσης πρέπει να πω ότι η νεολαία συμμετέχει στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών. Στα προγράμματα αυτά ελέγχει ότι θα πρέπει να έχουμε ε, περισσότερη υποστήριξη για την επαγγελματική εκπαίδευση στα πλαίσια του Λεωνάρδο. Στα πλαίσια του Λεωνάρδο φέτος τα 2 τρίτα των ποσών που δαπανίσαμε πήγαν για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και το 1 τρίτο για ανώτατη εκπαίδευση. Πράγμα που εξηγεί και το πρόβλημα που έχουν τα σχολεία, διότι φέτος δεν είχαν προτεραιότητα, διότι στο είπαν προτεραιότητα σε δύο, κατά δύο τρίτα δόθηκε στον επαγγελματική εκπαίδευση και τον τρίτο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτά ήθελα να πω. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Σα ευχαριστούμε πολύ για τι απαντήσει σα, για την παρουσίασή σα για όλε αυτέ τι πληροφορίε να σας ευχαριστήσω και όλους που συμμετείχατε στην σημαντικότατη αυτή συζήτηση. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μείνετε όσοι είστε συντονιστές στην αίθουσα αυτή, προκειμένου να συνεχίσουμε με τις συνεδρίες των συντονιστών.